Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω έχει, αρχίσει, έχει έρθει η ώρα συγγνώμη, να αρχίσουμε. Σημείο πρώτο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση του σχεδίου αυτή. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη χωρίς ε, τροποποιήσει. Και μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο σημείο Chairman's announcement. Ανακοινώση Προέδρου. Ανακοίνωση πρώτη. Για το θέμα των ε, γενετικά τροποποιημένων. Ναι. Στις 13 Ιανουαρίου ενέκρινε το Κοινοβούλιο μια πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και έχουμε το διορθωτικό κείμενο, το τελικό, μετά από γλωσσική επαλήθευση σε όλες τις γλώσσες, σύμφωνα με το άρθρο 231 εδάφιο 3 του κανονισμού. Το διορθωτικό έχει ε, σταλεί την Τετάρτη σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις μέχρι το τέλος, της σημερινή συνεδρίαση θα θεωρηθεί εγκεκριμένο το διορθωτικό και θα υποβληθεί αρμοδία στην Ολομέλεια στη Σύνοδο του Φεβρουαρίου. Δεύτερο. Το εργαστήριο για την δημόσια υγεία, για την αντίσταση στα αντιβιωτικά θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου, μία με τρεις, ε, εισηγητής είναι ο κ. Πεντητσίνη για το θέμα αυτό. Επόμενο θέμα. Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με συμμετοχή μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων για το ΠΟΠ 21 στο Παρίσι μέχρι το 2050, ο χάρτης και Ευρώπη ε, χωρίς ε, πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δευτέρα, 30 Μαρτίου το απόγευμα θα γίνει αυτό. Οι άτυπη. Το πρόγραμμα Life χτες ε, συνεδρίασε η άτυπη ομάδα και εξέλεξε τον κύριο Καπούτο και την κυρία Σουίτσα ως είναι μια ομάδα εργασία τη ΕΝΒΗ, εκεί συμμετέχουν ένα μέλος από κάθε πολιτική ομάδα, αλλά είναι δημόσιε συνεδριάση, Αν θέλετε και ενδιαφέρεστε μπορείτε να συμμετέχετε. Σήμερα η διερμηνία διατίθεται σε 22 γλώσσε. και συνήθως στο e-meeting έχετε όλα τα έγγραφα και ηλεκτρονικά της συνεδρίασης και επίσης η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται απευθεία από το διαδίκτυο. 22 Ιανουαρίου τι αποφάσισαν οι συντονιστέ. Έχει κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά το κείμενο με τι συστάσεις των συντονιστών. Αν δεν έχετε αντιρρήσει μπορεί να θεωρηθεί εγκρίθεν. Ωραία, μπορούμε να πάμε τώρα στο σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη που είναι οι ψηφοφορίε point on the vote, it is uh, Εκλογή συμπροέδρων της Ομάδας Εργασίας για την Υγεία. Στις 24 Ιουλίου οι συντονιστές αποφάσισαν να επανασυστήσουν την Ομάδα Εργασίας για την Υγεία μετά την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίασή τους στις 4 Δεκεμβρίου. Οι συμπροεδροί για την ομάδα Εργασίας για την Υγεία ε, θα εκλεγούν από τα μέλη της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Η προθεσμία για τις προτάσεις από τις πολιτικές ομάδες ορίστηκε για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 5 το απόγευμα. Έχουμε λάβει πέντε υποψηφιότητες. Γκούε, την κυρία Κίλονεν, η ΕΛΚ, Πέτερλε, η ΣΥΑΡ, τον κύριο Πιέκα, από τους Προσύνους, την κυρία Ριβαζή και από τους σοσιαλιστές την κυρία Γουίλμουτ. Πρέπει να ρωτήσω όλους τους υποψηφίους αν συμφωνούν ε, με την υποψηφιότητά τους. Και έχουμε λάβει από τον κύριο Πέτερλε, ο οποίος απουσιάζει, και από κάποιον άλλον, από την κυρία Ριβαζή επίσης, ένα mail που δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται την υποψηφιότητα. Οι υπόλοιποι, κυρία Κίλωνεν, συμφωνείτε, ναι. Ο κύριος Πιέκα, βεβαίως. Και η κυρία Βίλμουτ. Αποδέχεστε. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι σας έχουν διανεμηθεί ψήφο δέλτια. Παρακαλώ ελέγξτε αν έχετε λάβει όλοι το αντίστοιχα. Και πρέπει να σας ε, ενημερώσω ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της Επιτροπής και σε περίπτωση που απουσιάζουν μπορούν να αντικατασταθούν από αναπληρωτές σύμφωνα με τον κανονισμό. Ε, κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Μπορείτε να βάλετε σταυρό ε, για να ψηφίσετε στο όνομα που σας ενδιαφέρει και επίσης πρέπει να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να ψηφίσετε όποτε θέλετε και θα συλλέξουμε τα ψηφοδέλτια αμέσως μετά. Θα γίνει καταμέτρηση και στο τέλος της ψηφοφορίας, της ώρας ψηφοφορίας, θα σας ανακοινώσουμε το αποτελέσμα, γιατί πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Αν ψηφίσατε, μπορώ να ζητήσω λοιπόν να μαζέψουμε τα ψηφοδέλτια. Ε, the voting card. One minute to ένα λεπτό λοιπόν να περιμένουμε. going to go Okay, we can go... Καλώς μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Τις ψηφοφορίες δηλαδή για την απαλλαγή του 2013 του Γενικού Προϋπολογισμού θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία αμέσως. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 3. Με καταδιέρεση ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5 ψηφίζεται. I'm sorry, Mr. Sherman, but I ha I have... Συγγνώμη, δεν έχω φέρει την ε, κάρτα μαζί μου. Μπορώ να ψηφίζω δια ανατάσεως. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις Ας περάσουμε τώρα στην απαλλαγή για την υπηρεσία για τις φαρμακευτικές ουσίες. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τελική ψήφος ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτό. Περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Απαλλαγή για το ECDC. Ποιοι είναι υπέρ ε, του 1, τροπολογίας 1. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτό. Περνάμε στο 8. απαλλαγή για το 13 για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΣΑ. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε αμέσως τώρα στην τροπολογία 4. Κατά διέρεση ψήφος πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 5. Μια προφορική τροπολογία εδώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική. Οι σοσιαλιστές διαφωνούν. Αρκεί αυτό. Συνεπώς η προφορική τροπολογία δεν τίθεται σε ψηφοφορία και ψηφίζουμε τώρα την αρχική τροπολογία 5 χωρίς την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. Η τελική ψηφοφορία λοιπόν για την ΕΦΣΑ ηλεκτρονικά ψηφίζεται. Avete votato tutti. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας δεκτό το ψήφισμα. Περνάμε τώρα στο σημείο 9, απαλλαγή για το 13 για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών. Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 2, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ψήφος με ηλεκτρονικό τρόπο ψηφίζεται. Avete votato tutti, il voto όλοι πέρα της ψηφοφορία δεκτή η πρόταση. Τώρα περνάμε στο σημείο 10, απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ? κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 3 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 4 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραστη της ψηφοφορίας. Δεκτό. Περνάμε στο σημείο 11. Γνωμοδότηση του κυρίου Γραμματικάκη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εμενταμέντο 1. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 6. <laughs> Il voto è chiuso. Πέραση ψηφοφορίες Απερίφθη. γιατί η κυρία που δεν έχει την κάρτα ψήφισε κατά 33 με 33 συνεπώς απερίφθη. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Τροπολογία 8 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν απορρίπτεται. Τροπολογία 10 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τροπολογία 9 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τροπολογία 11 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τροπολογία 12 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 17 ψηφίζεται. Avete Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Τροπολογία τώρα 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 19 και 20 ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ. Εναντίον. Αποχές απερίφθη. 21. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 21. Ψηφίζεται. Il voto chiuso. ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 24. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 25. Ποιοι είναι υπέρ. Εναντίον αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 25. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη. 26. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 27 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική υπαριθμένα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 38 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 39 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 40. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τελική ψήφος ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Huh? Ε? Adesso abbiamo il... Τώρα έχουμε ηλεκτρονική ψήφο στην προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Στρατηγική για το Ινόπνευμα, το σημείο 12. Λοιπόν, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε ε, έναν επιπλέον από το FDD Πέρας της ψηφοφορίας δεκτή. Ομόφωνα. Θα πρέπει να ανακοινώσω τώρα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ομάδα εργασίας. 61 μέλη ψήφισαν, 19 ψήφοι για την κυρία Βιλμότ, 17 ψήφοι για τον κύριο Πέτερλε, 10 ψήφοι για την κυρία Ριβαζή, 7 ψήφοι για τον κύριο Πιέγκα, 5 για την κυρία Κιλόνεν και 3 λευκά ψηφοδέλτια. Αποτέλεσμα Έχουμε δύο εδώ εκλεγμένους, την κυρία Βιλμότ και τον κύριο Πέτερλε. Now we can go to the 13. Περνάμε τώρα στο 13. Το 13 της ημερήσιας διάταξης η στρατηγική για το ενόπνευμα και θα ξεκινήσω δίδοντας τον λόγο στον συνεισηγητή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τον κύριο Τσίριο. Grazie, grazie Presidente e un Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι εργάστηκαν αυτές τις τελευταίες εβδομάδες για τη σύνταξη του συγκεκριμένου σχεδίου. Πρόκειται για ένα θέμα θα έλεγα ευαίσθητο και σημαντικό ταυτόχρονα, το θέμα δηλαδή της στρατηγικής την οποία πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη για να μειώσει στο ελάχιστο ε, τις ζημίες οι οποίες προκαλούνται από την κατάχρηση των αλκοολούχων. Η πρόταση αυτή λοιπόν ψηφίσματος έχει βασιστεί σε ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες βασίζονται με τη σειρά τους στα στατιστικά στοιχεία τα οποία διαθέτουμε και σε επίπεδο ιστορικό αν θέλετε τα τελευταία χρόνια για τις ζημίες οι οποίες έχουν προκληθεί και σε επίπεδο απώλειας ανθρώπινης ζωής, σε επίπεδο υγείας, και φυσικά χωρίς να αγνοούμε και την οικονομική ζημία στα εθνικά συστήματα υγείας, ε, τα διάφορα κόστη γενικότερα. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για ενόπνευμα πάρα πολύ συχνά μιλάμε για καταστάσεις κοινωνικές ε, ε, με ιδιαίτερα τροτές κατηγορίες του πληθυσμού. Μιλάμε για κατάχρηση ενοπνεύματος από ανηλίκους, από ανθρώπους της ε, με κοινωνικά προβλήματα κτλ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό το οποίο έχει σημασία για να μπορέσει κανείς να εκφράσει τις απόψεις του είναι να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να διαφοροποιήσουμε τη δράση μας. Να μην θεωρήσουμε δηλαδή ότι η κατάσταση κατάχρησης του ινοπνεύματος είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο ακριβό τρόπο σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Εμείς ακούμε διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικά πλαίσια, πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά και γι' αυτό ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το ενόπνευμα οι κοινωνίες μας διαφοροποιείται και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να μην αντιπροτείνουμε μία συνταγή για την αντιμετώπιση του προβλήματος παντού. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν ε, ε, τις, τους τρόπους αντιμετώπισης και αντίληψης για το ενόπνευμα. Είναι διαφορετικό ε, να δει κανεί το τι αντιπροσωπεύει το κρασί σαν παράδειγμα στην περιοχή της Μεσογείου ενώ ε, με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζεται η κατανάλωση ποτών σε άλλα μέρη του κόσμου. Επίσης ε, υπάρχουν και διαφορετικές γαστρονομικές ε, καταβολές και παραδόσεις ε, στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης, στη Μεσόγειο κτλ. Μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Ένα από τα κομβικά σημεία λοιπόν του ψηφίσματος αυτού είναι η ικανότητα διαφοροποίησης της απάντησης. Μία ανάλυση λοιπόν για να είναι μια σωστή και συγκεκριμένη ανάλυση και η οποία να δείχνει με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται το ενόπνευμα και η κατανάλωση ενόπνευματος στα διάφορα κράτη-μέλη, είναι μια αντιμετώπιση η οποία θα έλεγα δεν θα πρέπει να στοχεύει μόνο στην δαιμονοποίηση και την απαγόρευση, αλλά στη σωστή εκπαίδευση, την εκπαίδευση στα σχολεία, την εκπαίδευση στην οικογένεια, ε, γιατί αυτό φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι να απαγορεύσουμε αλλά να ενημερώσουμε, να πληροφορήσουμε. Και αυτό είναι ένας από τους στόχους τους οποίους θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαν παράδειγμα η ετικετοθεσία, η σήμανση των αλκοολούχων προϊόντων, που θα έπρεπε να είναι κάτι το διαφορετικό από τις ετικέτες οι οποίες επιβάλλονται στα υπόλοιπα τρόφιμα. Αλλά ε, θα έπρεπε να κάνει τη διαφοροποίηση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον προηγούμενο Δεκέμβριο και από εκεί και πέρα θα βλέπαμε αν ε, αυτά τα οποία ισχύουν γενικότερα για τα τρόφιμα ισχύουν και για τα ίνοπνευματόδια. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια πολλαπλότητα, πολλαπλότητα καταναλωτών, μορφών κατανάλωσης, πολιτισμών γύρω από την κατανάλωση. Έχουμε το θέμα της σημασίας του σχολείου, της οικογένειας και δεν θα πρέπει να είμαστε άκαμπτοι σε σχέση ιδιαίτερα με τους νέους για τους οποίους η κατάσταση, η κατανάλωση του πνεύματος, δημιουργεί προβλήματα και τραύματα άμεσα. Και θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος και στην οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποιες εθνικές διαφορετικές απόψεις και ρυθμίσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει μηδενική ανοχή, δηλαδή η παρουσία υνοπνεύματος στο αίμα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το μηδέν, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει ένας διαφορετικός πολιτισμός γύρω από το θέμα αυτό, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί γύρω από αυτό και θα πρέπει να δούμε και το θέμα της υψηλής εθνιτότητας, θνησιμότητας, συγγνώμη, η οποία προκαλείται από την οδήγηση μετά από κατανάλωση νοπνεύματος. Μια τελευταία σκέψη τώρα. Η θέση μας είναι ε, όχι να θεωρήσουμε τη δυνατότητα μιας απλής καταδίκης σε πάση περιπτώσει των αλκοολούχων ουσιών όπως ακριβώς ε, ε, το έχουμε κάνει για τα προϊόντα καπνού. Αντίθετα, θα πρέπει με διαφορετικό τρόπο και με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε να δούμε και τις στατιστικές οι οποίες είναι αποκαλυπτικές εκεί όπου έχουν υιοθετηθεί κανόνες οι οποίοι έχουν αυξήσει την τιμή σαν παράδειγμα του υλοπνεύματος δεν έχει οδηγηθεί η κατάσταση στη μικρότερη κατανάλωση, στη μείωση της κατανάλωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρόκειται σε συγκεκριμένη περίπτωση για μια ισόρροπη πρόταση. Μια πρόταση και θα κλείσω εδώ η οποία έχει σαν στόχο να υιοθετήσει την σωστή πρακτική ε, της παράτασης ε, της λειτουργίας αυτού του φόρουμ έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητηθούν κάποια θέματα ε, και από πλευράς των χρηστών, των καταναλωτών και από την άλλη πλευρά των παραγωγών υπό τον έλεγχο των θεσμικών οργάνων. Αυτή η ομάδα εργασίας κατά κάποιο τρόπο έχει λειτουργήσει και νομίζω ότι πρόκειται για μια ορθή πρακτική την οποία θα πρέπει ε, της χρήσης, την χρήση της να τη διευρύνουμε. Η κυρία Βίλμοτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με στηρίξατε για να μπω σε αυτή την ομάδα που μόλις αποφασίστηκε. Χαίρομαι γιατί είχαμε ένα ψήφισμα στην προηγούμενη θητεία. Χαίρομαι που ξεκινήσαμε την ε, ενασχόληση με το θέμα αυτό, αλλά μετά ήρθαν οι εκλογές και δεν προλάβαμε. Σε αυτό το ψήφισμα τι ζητάμε. Μόνο και μόνο να υποβάλει νέα στρατηγική η Κομισιόν για το ενόπνευμα, για την ενοπνευματόδη. Η προηγούμενη έληξε το 2012 και ακόμη τίποτα. Η προηγούμενη στρατηγική βοήθησε να υπάρξει συνένεση στην Ευρώπη για το πώς να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που προκύπτουν από την ε, χρήση ενόπνευματος. Χρειαζόμαστε συνεργασία περισσότερη μεταξύ των κρατών μελών. Λοιπόν, μια νέα στρατηγική που να βασίζεται στην προηγούμενη. Για παράδειγμα, ίσως χρειάζονται περισσότεροι πόροι για την έρευνα, για τη βλάβη που προκαλεί η κατανάλωση υνοπνευματοδών, να δούμε ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν, να δούμε αν θα μπορούσαν ε, να υπάρχουν ελάχιστε τιμές. Επίσης και οι κανόνες σήμανσης. Όταν συζητούσαμε την οδηγία για την πληροφορία τροφίμων είχαμε εξαιρέσει τα ενοπνευματόδη. Γιατί όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από άλλα τρόφιμα. Ήμουν κατά αυτής τη εξαίρεση. όμως η Κομισιόν τότε είχε πει ότι θα υποβάλει έκθεση για να επεκταθούν και στα ενοπνευματόδη μέχρι τον ε, παρελθόντα Δεκέμβριο να επεκταθεί και στα ενοπνευματόδη η οδηγία αυτή. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Φυσικά η σήμανση θα πρέπει να λέει ότι είναι επικίνδυνο να οδηγεί υπό την επίρρεια ορματοδών, ε, όταν είναι κανεί ανήλικος ή όταν είναι έγκυος τι κίνδυνοι προκύπτουν από την κατανάλωση νοηματοδόνα, αλλά πρέπει να έχουμε και για τη θερμιδική αξία πληροφορίες. Πολλοί λένε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πολλοί παραγωγοί ήδη δίνουν αυτή την πληροφορία. Δεν είναι άρα και τόσο δύσκολο. Θέλω λοιπόν να είμαι απόλυτα σαφής, γιατί ξέρω ότι πολλοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για αυτό το θέμα. Όχι, δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε τον πνευματόδη. Δεν πρόκειται να εμποδίσουμε την κατανάλωση, ούτε να αλλάξουμε τις συνήθειες ενός ή άλλου λαού, ούτε θέλουμε να καταγγείλουμε αυτούς που ε, πίνουν πνευματόδη, ούτε να σταματήσουμε την παραγωγή ε, ίνου από διάφορες χώρες. Και εγώ πίνω λίγο κρασί. Αλλά είναι θέμα δημόσιας υγείας. Διότι τα ενοβλεματόδη είναι το τρίτο αίτιο ε, ασθενειών στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να προληφθούν. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στους καταναλωτές ε, τις πληροφορίες ε, που χρειάζονται για να κάνουν τις σωστές επιλογές. Αν θέλουμε να μειώσουμε τη ζημία από τα εινοπνευματόδη πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα μέσω ψηφίσματος προς την Επιτροπή ότι πρέπει να αναλάβει δράση για το θέμα αυτό και ότι είναι επιτέλους ε, ε, η ώρα να υποβάλει και μάλιστα έχει καθυστερήσει να υποβάλει προτάσεις για αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φάρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους που συνεργάστηκαν για να καταλήξουν σε αυτή την πρόταση. Η κατάχρηση πινοπνευματοδών ε, προκαλεί πολλές ασθένειες, πρόωρους θανάτους ε, και έχει επίπτωση και στην οικονομία. Αρνητική. 150 εκατομμύρια το χρόνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν ήδη από το 2012 την προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό αλλά είμαστε ήδη το 2015 και θα πρέπει να μας υποβάλει νέες προτάσεις για την αντιμετώπιση πνευματοδών, διότι η κατανάλωσή τους εξακολουθεί να είναι ουσιώδης κίνδυνος για τις ε, κοινωνίες μας και από οικονομική άποψη και από κοινωνική άποψη. Υπάρχουν θέματα που νομίζω ότι είναι βασικά για το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε σαφή διαχωρισμό μεταξύ της ε, λογικής κατανάλωσης και της υπερβολικής κατανάλωσης λαμβάνοντα υπόψη και τις διαφορές ε, ε, στις διάφορες χώρες και τις διαφορές στο βαθμό ε, στις διαφορές στο βαθμό που είναι ευάλωτα διάφορα τμήματα του πληθυσμού δηλαδή η ηλικία κατά την οποία αρχίζει κανείς να πίνει κτλ. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν και μελέτες για το θέμα αυτό για, τα, για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης υλοβρομάτοδων, ούτως ώστε να είναι πιο επιστημονικές οι προτάσεις μας και να βελτιώσουμε φυσικά κάθε μέτρο που θα ευνοήσει τη σωστή πρακτική, τις σωστές πρακτικές, βασιζόμενοι σε όλα τα μέτρα που έχουμε υιοθετήσει μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει συντονισμός ε, μεταξύ κρατών μελών, κυρίως όσον αφορά τη σήμανση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει φραγμούς και πρέπει να το αποφύγουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση ψηφίσματος είναι καλή, ισορροπημένη, όπως έχει ήδη υποθεί και ήθελα να προσθέσω ότι ούτε πρέπει, ούτε είναι δυνατό να αντιμετωπίσουμε τα ενοπνευματόδη όπως ε, τα προϊόντα καπνού όπως είπε και η προηγούμενη ε, ομιλήτρια, γιατί ένα ποτήρι κρασί, ιδίως αν είναι κόκκινο, ε, μπορεί να ωφελήσει. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω ε, στις ε, ερωτήσεις σας. Εμείς οι συνζήτες είμαστε στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε τα κρασιά. Υπάρχουν πορτογαλικά καλά κρασιά, αλλά υπάρχουν και πολύ καλά ε, κρασιά στη χώρα μου. Κυρία Γκίρινγκ. Ε, μπορεί να σε εκπλήξει, αλλά έχουμε κρασιά και στην ε, Αγγλία. Έχουμε κυρίως άσπρο βέβαια, αλλά είναι πολύ καλό. Ε, εκπροσωπώ τον συνάδελφο Πρέτσελ, ο οποίος ε, έφυγε. Συμφωνούμε ότι είναι θέμα τα ενοπνευματόδη είναι είναι το τρίτο αίτιο ε, ασθενειών που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και μας ενδιαφέρει ως θέμα δημόσιας υγείας, έχει να κάνει και με την παχυσαρκία και τον διαβήτη. Όλα αυτά συνδέονται με την κατανάλωση ινοπλεύματος. Αλλά μας ενδιαφέρει και κάτι που ήδη υπόθηκε. Με συγχωρείτε που λέω ότι είναι θέμα πολιτισμού. Υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές. Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο παράγεται, ε, πωλείται και καταναλώνεται. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Άρα δεν είναι δυνατόν ε, να νομοθετήσουμε ένα μέτρο για όλους. Τα κράτη-μέλη πρέπει να πάρουν ε, τις κατάλληλες αποφάσεις και γιατί να μην θεωρήσουμε ότι μπορούν να λάβουν τις, τις πιο κατάλληλες για τη χώρα τους. Άρα δεν είναι ρόλος μας εμείς να τα αποφασίσουμε όλα αυτά, αλλά μπορούμε να ε, αποφασίσουμε για τη σήμανση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις θερμίδες που περιέχει. Γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τους νέους που πίνουν υπερβολικά, βγαίνουν έξω το βράδυ, γιατί οι νέοι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για το σώμα τους, άρα μπορεί να βοηθήσει να μην πίνουν πολύ. Γιατί το θέμα δεν είναι η ποσότητα πνεύματο. Ξέρουμε ότι μειώνει τη μέση κατανάλωση, αλλά είναι ο τρόπο κατανάλωση. Πού πίνουμε. Και αυτό το φαινόμενο του να πίνει κανεί πολλά ένα βράδυ, ξέρω ότι θεωρείται από πολλού ε, βρετανικό φαινόμενο, βρετανική ασθένεια. Και δεν μου αρέσει που ακούγεται αυτό για τη χώρα μου, αλλά υπάρχει στη χώρα μου. Άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε νομίζω θα βοηθούσε. Αλλά φυσικά δεν θέλουμε να είναι υπερβολικά βαριά και λεπτομεριακή η νομοθεσία γι' αυτό, γιατί πολλές φορές όλοι θεωρούν, ορισμένοι θεωρούν ότι ενόπνευμα και τσιγάρο είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Μία λογική, μετρημένη κατανάλωση ενόπνευματος μπορεί να είναι και εποφελής Αλλά όποιος πίνει υπερβολικά και μάλιστα προσπαθεί να μεθύσει γρήγορα βγαίνοντας το βράδυ, φυσικά δεν κάνει καλά. Αλλά δεν πρέπει να είναι υπερβολικά παρεμβατική η νομοθεσία μας. Ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να έχουμε ελάχιστες τιμές ανά ενότητα υνοπνεύματος. Δεν ξέρω όμως αν αυτός είναι ο καλύτερος μακροχρόνιος τρόπος για να περιορίσουμε την κατανάλωση. Ξέρω ότι έχει επιχειρηθεί σε ορισμένα τμήματα της ενός, αλλά δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της κατανάλωσης, άρα προσεκτικά να το δούμε αλλά το βασικό είναι η στρατηγική μας να αντιμετωπίσει τα θέματα με ευαίσθητο και λελογισμένο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό στην ουσία βασίζεται σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προσέξει και να το αντιμετωπίσει. Η στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε ήδη από το 2006 έχει λήξει από το 2012. Ε, πήρα μέρος στην ε, σύνταξη αυτής της πρότασης μαζί με άλλους συναδέλφους ε, βασισμένος στην ανάγκη να υπάρχει περιορισμένη χρήση και κατανάλωση των συγκεκριμένων ουσιών έτσι ώστε να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στην χρήση και στην κατάκριση. Η καταπολέμηση λοιπόν του των ενοπνευματοδών θα πρέπει να αναγνωρίζει αν θέλετε κάποιες πραγματικότητες. Ε, στους πληθυσμούς άνω των 15 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει φτάσει το 10,77 λίτρα. Στην Ιταλία για να το παραλληλήσω με την Πορτογαλία, έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό και καταναλώνουμε 6,94 λίτρα κατέτος κατά κεφαλήν. Και παρόλα αυτά είμαστε μεγάλη παραγωγός χώρα. Και υπάρχει και μία μείωση γενικότερα, μία τάσικα μείωση της κατανάλωσης εδώ και πολλά χρόνια. Στις εξαγωγές μας ε, κυρίως εξάγουμε ε, κρασί, μούστο, είναι ποτά με υψηλή, υψηλό βαθμό υνοπνεύματος που παράγονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για να μην πω από πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε τις επιβλαβείς συνέπειες του ε, προϊόντος χωρίς να βλάψουμε τις τοπικές παραγωγές, γιατί έχουμε εμπειρίες διαφορετικές από ό,τι στο βορρά της στην Ευρώπη και μπορούμε έτσι να συνεισφέρουμε με επικοδομητικό τρόπο στη δημιουργία μιας σωστής στρατηγικής. Δεν ξέρω αν η κυρία Κονέτσνα θέλει το λόγο. Έχετε το λόγο κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω από πλευρά της ομάδας μου ότι μας αρέσει το κείμενο αυτό γιατί τονίζει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Συζητάμε διάφορες ε, εξαρτήσεις συχνά. Αλλά... Α, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη διερμηνία, λέει ο πρόεδρος. Στα γαλλικά. Okay, probably we can... Okay, thank you. Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία άλλη ουσία που να οδηγεί για παράδειγμα σε διάλυση οικογενειών, ε, βία εντός των οικογενειών και εκτός. Υπάρχουν τρομερές, τρομερές κοινωνικές επιπτώσεις από την ε, κατάχρηση νοπνεύματος δεν μπορεί να συγκριθεί από αυτή την άποψη με το καπνό. Ο καπνός δεν προκαλεί βία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να περιορίσουμε σοβαρά την ε, κατανάλωση πνεύματος, αλλά πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Διότι σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν καθόλου περιορισμοί για την κατανάλωση νοπνευματοδών. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να το τονίσω. Και έχει να κάνει, για παράδειγμα, με τη διαφήμιση. Η διαφήμιση νοπνευματοδών. Αυτό δεν είναι θέμα παραδόσεων ε, καμιάς κοινωνίας. Αλλά αν τα παιδιά βλέπουν συνέχεια διαφημίσεις από πολύ μικρά στην τηλεόραση ότι α, το να πίνεις ε, είναι φυσιολογικό τότε ε, πιο εύκολα θα αρχίσουν να πίνουν και εκείνα. Θα θεωρήσουν ακριβώς ότι είναι φυσιολογικό. Άρα πώς θα περιορίσουμε την κατανάλωση έτσι. Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να πίνουν ε, λογικά, πολύ εύκολα μπορεί να γίνουν αλκοολικοί. Γιατί πρέπει να διαφημίζουμε τα ενοπνευματώδη, γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε ε, τέτοιου τύπου παραγωγού. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Κάτι που επίση αναφέρεται εν μέρει τουλάχιστον στο κείμενο. Στο 22 λέτε λέτε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε και να εφαρμόσουμε στρατηγικές για ένα υγιή τρόπο, τρόπο ζωής μέσω αθλητισμού και υγιεινών συνηθιών διασκέδασης. Σκεφτείτε πόσα για παράδειγμα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις έχουν ως χορηγούς εταιρείε συνοπνευματοδών οι διαφημίσεις για ενοπνευματώδη ε, είναι πανταχού παρούσες όταν βλέπει κανείς ε, διάφορες ε, αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες. Έτσι μαθαίνουμε τα παιδιά μας. Έτσι τα μαθαίνουμε ότι είναι φυσιολογική η κατανάλωση ενοπνευματώδων. Καλά εντάξει δεν είναι κακό να πιει κανείς ένα ποτήρι πορτογαλικό, ισπανικό, ιταλικό ή τσεχικό κρασί. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κρίνουν. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τα παιδιά να θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό να πίνει κανείς ενόπνευμα. Άρα το θέμα είναι η διαφήμιση. Αυτό θέλω να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτό να εστιάσουμε. Δεν χρειάζεται. Και δεν νομίζω ότι προσθέτει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζώμα. Ναι. Η ε, απαγόρευση των διαφημίσεων βέβαια είναι ένα θέμα πάντα αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ διαφωνώ. Η διαφήμιση για το ενόπνευμα απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους, αλλά και η χορηγία είναι σημαντική. Για αθλητικούς συλλόγους, ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ήπεθρο είναι σημαντικό. Δεν έχουν σπόνσορες, δεν έχουν ε, επιδοτήσεις και στη Γερμανία πολλές διθοποιίες τοπικές υποστηρίζουν τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και δεν νομίζω ότι θα πρέπει ε, καταρχήν να απαγορευθούν. Ε, δεν μας αρέσει αυτό. Ε, για το σχέδιο ψηφίσματος γενικά μου αρέσει πολύ αλλά θέλω να διορθώσω κάτι στο σημείο, στην αιτιολογική σκέψη μάλλον ο Μικρόν που λέει ότι ε, ο κανονισμός για τα τρόφιμα έχει εξαιρέσει το ενόπνευμα. Δεν ισχύει αυτό. Βεβαίως ρυθμίζεται με τον κανονισμό αυτό. Θα πρέπει να αναφέρεται ο αλκοολικός βαθμός ε, και υπάρχουν και άλλες υποχρεωτικές αναφορές τα ενοπνευματόδη μόνο εξαιρούνται από τις θερμίδες και από το κατάλογο των συστατικών. Και αυτό μάλιστα θα είναι μεταβατική ρύθμιση πιστεύω διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φέρει μια έκθεση και μάλιστα ε, σωστά αναφέρομαι ότι έπρεπε ήδη να έχει έρθει από το Δεκέμβριο. Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Αν μιλάμε για σήμανση ως προς τις θερμίδες και τη θρεπτική αξία είναι κάτι στο οποίο έχω επιφυλάξει και το έχω ξαναπεί και θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Ε, η σήμανση που επιβάλλει ο κανονισμός για τις δείκτες ε, προβλέπει τη μονάδα μέτρησης 100 ε, ml ή 100 γραμμάρια. Για την πύρα και το κρασί αυτό είναι εντάξει, αλλά για εινοπνευματόδη υψηλού αλκοολικού βαθμού είναι επικίνδυνο γιατί υπάρχουν πολίτες που θεωρούν ότι 100 ml ρακή ας πούμε ή σναπς είναι εντάξει αν θεωρηθεί θερμίδα και ότι μπορούν να πίνουν τόσο και μάλιστα άμα το λέει και ο κανονισμός είμαστε καλυμμένοι. Όχι, αυτό θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε μήπως να το σταθμίσουμε καλύτερα γιατί είναι και επικίνδυνο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου χρόνια τώρα να τα λέω αυτά. Ε, άλλα θέματα από την έκθεση Πιστεύω ότι η αναφορά τη ελάχιστη τιμή θα πρέπει να διαγραφεί. Μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία καθόλου. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να παραπέμπουμε σε θετικέ εμπειρίε. Κατά τα άλλα, η φορολογική νομοθεσία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε και θα πρέπει να παραμείνει φυσικά κατά την άποψή μου. Εκεί τα κράτη-μέλη έχουν ήδη βρει σωστές ρυθμίσεις και σε ό,τι αφορά την προστασία των ανελίκων από την υπερβολική κατανάλωση νοπνευματοδών, ιδιαίτερα τα προϊόντα που ονομάζονται αλκοπόψ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ελάχιστες τιμές ε, στα ενοπνευματώδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, συνολικά θα πρέπει να δούμε ότι δεν έχουν θέση στην έκθεση αυτή στοιχεία παγκόσμια ε, γενικά, αλλά παρακαλώ συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση εργαζόμαστε. Äh, και θέλω να σας πω επίσης ότι, εξ όσο γνωρίζω, οι 10.000 νεκροί από τροχέα που ε, ανάγονται στο αλκοόλ δεν ισχύει αυτό, έχει αλλάξει. Έχει μειωθεί στο μισό ο αριθμό των θυμάτων και έχουν φτάσει τις 5.000 πλέον. Αυτό χρειάζεται απόδειξη. Τώρα βέβαια και 5.000 και ένας έστω να είναι, είναι ε, ένας θάνατος ε, ε, που πρέπει να αποτρέπεται. Για τις προειδοποίησεις τώρα που αναφέρθηκαν στη συζήτηση, υπάρχουν ε, στα κράτη-μέλη σχετικές ρυθμίσει και δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να αφαιθεί αυτό και να ξεκολουθήσει να είναι στα χέρια των κρατών μέλων. Έχω κι εγώ επιφυλάξεις. Τι νόημα έχουν οι προειδοποίησεις πάνω στη φιάλη. Γιατί δεν το πίνεις από το μπουκάλι κάθε φορά το αλκοόλ. Δηλαδή, άμα έχει φτάσει να πίνει από το μπουκάλι, είσαι χαμένο έτσι κι αλλιώ. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφέρεται κάτι ε, στη φιάλη. Για τα παιδιά το έχουμε ξαναπεί να μην πίνουν αλκοόλ, αλλά το έχουμε ε, ξαναπεί αυτό ότι είναι θέμα γιατρών και ε, του υγειονομικού προσωπικού να το χειρίζεται. Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Τώρα προειδοποίηση πάνω στη φιάλη είναι αργά. Ε, θέλω να επισημάνω επίσης μια αντίφαση. Από τη μια λέει το σχέδιο ψηφίσματος ότι η στρατηγική μέχρι τώρα για την ε, κατάξυση του αλκοόλ ήταν πάρα πολύ ε, αποτελεσματική και από την άλλη ζητάει καινούρια. Για ποιο λόγο ε, υπάρχει τέτοια ανάγκη, άμα είναι επιτυχής και καλή η παλιά και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι λειτουργεί, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα κράτη-μέλη προς το ίδιο τους το συμφέρον δηλαδή τελικά και για να κάνουν και οικονομίες δεν μπορούν στο σύστημα υγείας και στο κοινωνικό σύστημα προστασίας να έχουν μια καλή πολιτική για την κατανάλωση αλκοόλ. Δεν ξέρω, στο ψήφισμα βλέπω αυτή την αντίφαση και με προβληματίζει. Ε, θα ήθελα να το ξανακοιτάξουμε. Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε αντιφάσεις μέσα σε ψηφίσματα. Και ένα τελευταίο, χαίρομαι πάρα πολύ που τονίστηκε από συναδέλφους εδώ ότι δεν μπορεί κανείς να βάλει όλα τα κράτη-μέλη στο ίδιο τσουβάλι Υπάρχουν διαφορετικά ήθη, έθιμα, συνήθειες, καταβολές, παραδόσεις. Ε, ακόμα και οι ε, αφορμές ή οι ε, ευκαιρίες που έχει καθένας να καταναλώνει αλκοόλ διαφέρουν. Δεν είναι όλοι οι πολίτες της Ένωσης το ίδιο. Ούτε θα πρέπει κάπως να προσπαθήσουμε να χαλιναγωγήσουμε όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο. Αυτό θα στείλει τους ε, Ευρωπαίους στην αγκαλιά των ε, λαϊκιστών της δεξιάς, πράγμα που δεν θέλει κανείς από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπότα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα πολύ άσχημα στατιστικά στοιχεία τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Μας δείχνουν με ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει νέα μέτρα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία συνδέονται με την κατανάλωση ινοπνεύματος από τους εργαζομένους Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ πηγαίνει στις, στη μετρίαση των συνεπειών της υπερβολικής κατανάλωσης συνοπνεύματος. Απαιτείται λοιπόν να έχουμε το πολιτικό θάρρος και να πούμε ότι οι καταναλωτές, ιδιαίτερα οι νέοι, έχουν μεγαλύτερη σημασία από ότι τα κέρδη και από ότι το κόστος της αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Το σηκώτη μιας γυναίκας ε, ε, επεξεργάζεται το ενόπνευμα τρεις φορές πιο αργά από ότι το ανδρικό σηκώτη και αυτό δείχνει ότι η γυναίκα μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από το ενόπνευμα πολύ πιο εύκολα από τον άνδρα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Σαν παράδειγμα βλέπουμε ότι η κατανάλωση νοπνεύματος είναι υψηλότερη στις πλούσιες χώρες και όχι τόσο στις φτωχές. Όμως οι πληθυσμοί των φτωχών χωρών υποφέρουν περισσότερο από την υπερβολική κατανάλωση, από την κατάχρηση. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα στρατηγική το ταχύτερο δυνατόν. Έτσι θα προετοιμάσουμε τον τρόπο ε, για μια καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος και να ε, εμποδίσουμε τους πολίτες μας ε, να κάνουν καταχρήση. Κατά στον, ε, του ίνοπνεύματος. Υπάρχουν επίσης και άλλα προβλήματα σε σχέση με την επισήμανση των προϊόντων, την ετικετοθεσία των προϊόντων και την ανταλλαγή των, των σωστών πρακτικών. Ευχαριστώ Ντελέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι μια καλή βάση εργασίας. Πρέπει να υπογραμμίσουμε κάτι το οποίο έγινε και από αρκετούς άλλους συναδέλφους, το ότι η κατανάλωση πνεύματος διαφέρει ιδιαίτερα από τη μία χώρα στην άλλη. Διαφορετικά συνήθεια, διαφορετικό ιστορικό αν θέλετε. Υπάρχουν τρία σημεία στα οποία θα σταθώ και πρέπει να τα προσέξουμε όλοι. Το πρώτο σημείο βρίσκεται στην παράγραφο 7. Είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Είναι η έννοια η οποία αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτή την έννοια μέσω σωστότερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης του καταναλωτή. Το δεύτερο σημείο είναι στην παράγραφο 26 Εκεί υπογραμμίζουμε το ότι θα πρέπει να στηρίξουμε ε, τα προβλήματα όπως ε, η πώληση παρανόμου εινοπνεύματος ε, ή κάποια προϊόντα τα οποία είναι ψευδεπίγραφα, δεν είναι τα γνήσια προϊόντα. Και τα νοθευμένα προϊόντα επίσης. Και το θέμα εδώ δεν είναι ότι έχουμε να κάνουμε με αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με αρμοδιότητες των κρατών μελών. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Στη Γαλλία έχουμε τον νόμο ΕΒΑΝ και γι' αυτό κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει τις δικές του εμπολείς ευθύνες. Ε, μια πρόταση ελάχιστης τιμής, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό γιατί στην ουσία επιβάλλουμε την εξέταση του θέματος μόνο μέσω της προβληματικής του κόστους. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κοινωνική σύγκληση, δεν υπάρχει δημοσιονομική σύγκληση, κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες αν θέλαμε να δημιουργήσουμε μια σωστή τιμολόγηση των αλκοολούχων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκροστέτ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι ε, πρόβλημα δημόσιας υγείας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά εγώ ακούγοντας όλους τους συναδέλφους θεωρώ ότι προς Θεού μην αρχίσει τώρα να νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλές οι συστάσεις, μπορεί να συστήνει διάφορα πράγματα στα κράτη-μέλη ως προς την πρόληψη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι πραγματικά η ε, ουσία και ε, στους νέους, τους, ε, στα παιδιά πριν από την εφηφική ηλικία. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες πολιτών που μπορεί να είναι πιο ευάλωτε ομάδε. Και αυτοί είναι οι ανήλικοι, οι νέοι, που είναι όλο και πιο μικροί στην ηλικία, που οι νοπνευματόδοι για να φτάσουν σε ένα επίπεδο ε, εφορίας που καταλήγουν σε ε, απώλεια της συνείδησης. Και αυτός γίνεται στόχος να πιείς, να μεθύσεις μέχρι να μείνεις ανέστητος. Και ο πρώτος ε, που θα λιποθυμήσει κερδίζει. Ε, ε αυτό δεν χρειάζεται ε, ρύθμιση αλλά συστάσεις για να υπάρξει πραγματικά πρόληψη που να έχει γίνει με πάρα πολύ καλό τρόπο σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού που είναι όλο και πιο νεαρότερη σε ηλικία παντού και στις έγκυες εάν το υγειονομικό προσωπικό δεν είναι σε θέση να εξηγήσει σε μια έγκυο γυναίκα τους κινδύνους της κατανάλωσης συνοπνεύματος για το ε, παιδί της, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και εκεί συστάσεις χρειάζονται όμως για να υπάρχει πρόληψη στα κράτη-μέλη και να εξηγούμε τις συνέπειες στην ανάπτυξη του εμβρίου, στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του κτλ. Όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι θα ήθελα και εγώ να κάνω μια διάκριση εδώ ανάμεσα στην λελογισμένη, ε, περιορισμένη μετριοπαθή κατανάλωση του υνοπνεύματος. Ε, ας πούμε όταν ε, πίνεις ένα ποτήρι πάρα πολύ καλό αλλά καλό κρασί και ένα ε, είναι απόλαυση αυτό ε, και όχι απλώς να πιείς ένα οποιοδήποτε ενόπνευμα για να μεθύσεις για την ε, σήμαση τώρα και τις ετικέτες έχουμε ήδη βάλει πάρα πολλά πράγματα στις ετικέτες Ας πούμε, κοιτάξτε τα μπουκάλια του κρασιού. Εγώ είμαι από μια χώρα ε, εγνωσμένης ε, και εφημισμένης ε, ε παραγωγή, παραγωγής και ξέρω ότι όσο περισσότερο φορτώνει στην ετικέτα τόσο λιγότερο τη διαβάζουν. Και έχει σημασία πάρα πολύ να πούμε αντιθέτως ότι η υπερβολική κατανάλωση πνεύματος είναι επικίνδυνη. Αλλά σταματήσουμε να επιβάλλουμε στους αμπελουργούς μας ετικέτες. Αν βάλουμε όλα αυτά που ζητούν ορισμένοι στην ετικέτα θα ε, ε, κάλυπτε όλη τη φιάλη. Δεν θα βλέπεις ούτε προέλευση ούτε τίποτα. Για την ελάχιστη τιμή, την ενιαία κτλ. Και αυτό είναι μια ε, ιδέα που μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως καλή αλλά δεν είναι ενισχύεται το λαθρεμπόριο με αυτόν τον τρόπο και οι καταναλωτές θα ε, ψάχνουν πηγές πολύ πιο επισφαλείς και ανεξέλεγκτες για να προμηθεύονται τα ενοπνευματοδήποτα, πράγμα που θα έχει επιπτώσεις και στους μηχανισμούς της αγοράς. Βεβαίως, το Ευρωπαϊκό Φόρμ για το Ενόπνευμα και την Υγεία έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν αντιλέγω, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στη Γαλλία, και τα είπε η συνάδελφος Ντελαέ, έχουμε μια ρύθμιση πάρα πολύ αυστηρή, ε, απαγορεύεται η διαφήμιση, απαγορεύεται η χρήση στους αθλητικούς χώρους. Αυτά ισχύουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά κυρίως να ενημερώνουμε και πρόληψη ε, στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγιούζου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ με όλους ε, και όλους όσους είπαν τόσα ενδιαφέροντα πράγματα στις παρεμβάσεις τους. Εγώ δεν είμαι κατά τον έχουμε στρατηγική για το ενόπνευμα, αλλά αν λειτουργήσε ε, η προηγούμενη, με μικρές μετατροπές θα μπορούσε να συνεχιστεί. Το θέμα της ουσίας είναι ότι δεν μπορούμε εμεί από εδώ να λύσουμε τα προβλήματα ορισμένων περιοχών σε ορισμένες χώρες. Η Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικούς τρόπους, μορφές κατανάλωσης συνοπληματοδών. Στο Νότο, για παράδειγμα, καταναλώνεται με κοινωνικό τρόπο και συνήθως με τρόφιμα το ενόπνευμα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με άλλες συνήθειες όπου Παρασκευή ε, βράδυ ή Σάββατο βράδυ πίνουν μέχρι να πέσουν εξαιρεί. Αυτό δεν συμβαίνει στον Νότο. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα μέτρο για όλους. Δεν μπορούμε να κατευθύνουμε και να καθορίζουμε τη ζωή όλων των ε, πολιτών μας. Τώρα για τη σήμανση. Συμφωνεί, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν στην ετικέτα. Βεβαίως οι αλλεργίες, η περιεκτικότητα κατόγκωση, ενόπνευμα και όλοι ξέρουν ότι παχαίνει το ενοπνευματόδες, ότι έχει ε, θερμίδες και όλοι ξέρουν, όλοι το ξέρουν αυτό, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσουμε. Όλοι όσοι πίνουν το ξέρουν. Λοιπόν, είναι ούτως άλλως και θέμα επικουρικότητα, γιατί ο καθένα έχει τα προβλήματά του στη χώρα του. Στην Ισπανία έχουμε πολύ αυστηρές ρυθμίσεις για το ενόπνευμα. Είναι περιορισμένη και η διαφήμιση και η πώληση. Είναι τρομερά αυστηρός ο κώδικας οδική κυκλοφορία. Όποιον πιάσουν με ένα ποτήρι παραπάνω πληρώνει τρομερά ποσά και του παίρνουν και το δίπλωμα. Έχουν γίνει όλα αυτά. Αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στη χώρα κάποιου άλλου, α το αντιμετωπίσει. Δεν χρειάζεται ομοιομορφία για όλου. Και για τι τιμέ βεβαίω, βεβαίω, οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται να παρέμβουμε. Δεν θα βοηθούσε να παρέμβουμε στην τιμή. Και για την Ισπανία υπάρχουν επιπτώσει γιατί έχουμε πολύ καλές διαφημιστικές εκστρατείες για την υπεύθυνη κατανάλωση του αυτό είναι το βασικά ε, σημαντικό, να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές. Έχει να κάνει περισσότερο με τους λόγους για τους οποίους πίνουμε, όχι με τις επιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε το κοινό για την υπεύθυνη κατανάλωση. Οτιδήποτε άλλο, όχι μόνο δεν είναι σωστό, αλλά μπορεί να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Ντόρφμαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές διότι πράγματι έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν υπογραμμίσει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην χρήση και την κατάχρηση. Αυτό είναι αυτό που έχει σημασία γιατί τα αλκοολούχα είναι τμήμα του πολιτισμού μας και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι παίζουν και σημαντικό οικονομικό ρόλο ιδιαίτερα σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης, ε, της Ευρωπαϊκής Υπέθρου. Έχουμε περιοχές της Υπέθρου στη χώρα μας που ζουν αποκλειστικά από την παραγωγή νοπνευματοδών, ιδιαίτερως κρασιού και από τις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες όπου έχουν και οικονομικό βάρος οι εξαγωγές αυτές των αλκοολούχων. Αυτό δεν κρύβει το ότι υπάρχει επίση η κατάχρηση και υπάρχει και εξάρτηση. Είναι μια ουσία η οποία προκαλεί εξαρτήσεις και οι εξαρτήσεις είναι ασθένειες. Και αναφέρομαι τώρα στις έγκυες. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν γνωρίζουν στην Ευρώπη τουλάχιστον ότι κατά τη διάρκεια της ε, της περίοδου αυτής δεν θα πρέπει να πίνουν υνοπνευματόδη. Και πράγματι είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό, φαίνεται και στα μέσα ενημέρωσης με τους διάσημους οι οποίοι ε, όταν πηγαίνουν σε δεξιώσεις δεν πίνουν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικό, κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι εξαρτημένες ε, μένουν έγκυες και δεν καταφέρνουν να σταματήσουν την εξάρτησή τους και αυτό έχει τρομερές συνέπειες στα άτυχα παιδιά. Εδώ είναι το πρόβλημά μας, πρέπει αυτές τις γυναίκες να τις βοηθήσουμε, να τις συνοδεύσουμε ε, ιατρικά, γιατί εδώ δεν είναι θέμα ενημέρωσης, είναι ιατρικό πρόβλημα και το είπε και ο κύριος Πεντιτσίνη, θα πρέπει να δούμε τη συνολική κατανάλωση του αλκοόλ ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπει κανείς ε, ενδιαφέροντα πράγματα σε μια χώρα σαν την Ιταλία, όπου υπάρχει μια μακρά παράδοση ινοπαραγωγής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν και άλλες μορφές κατανάλωσης. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με λιγότερο από ε, ατομική κατανάλωση κατέτος κάτω των 7 λίτρων. Πολύ λιγότερα, ε, πολύ μικρότερη κατανάλωση από χώρες ε, με πολύ μικρότερη παραγωγή υνοπνευματοδών από την Ιταλία, την Ισπανία κτλ. <coughs> Λοιπόν, ε, και μάλιστα πρώτες στην κατανάλωση είναι και χώρες οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν ε, τη λογική της απαγόρευσης ε, σαν βασικό μέσο για την αποτροπή της κατάχρησης συνοπνευματοδών. Αυτό δείχνει νομίζω ότι το θέμα της τιμολόγησης, της ελάχιστης τιμολόγησης ή της υψηλής τιμολόγησης δεν είναι κάτι το οποίο βοηθά. Όλα αυτά θα πρέπει να βασιστούν λοιπόν στο τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να τα διορθώσουμε, θα πρέπει να βασιστούμε επίσης σε αυτά τα οποία τώρα κάνουμε. Υπάρχει άλλωστε και το πρόγραμμα Wine in Moderation, το οποίο ο παραγωγικός τομέας εφαρμόζει γιατί ο ίδιος ο τομέας ε, θέλει να υπάρχει μέτρια κατανάλωση γιατί βαχυπρόθεσμα η υπερβολική κατανάλωση είναι κάτι το καλό για τους παραγωγούς αλλά μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν είναι κάτι το καλό ούτε για τους παραγωγούς. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια σωστή ισορροπία για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την υπερβολική κατανάλωση. Herbert. Σας ευχαριστώ. Γκαρντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω εδώ, πολλά ακούστηκαν. Ένα πράγμα νομίζω πρέπει να υπογραμμίσω, το οποίο το είπε και πάρα πολύ σωστά η κυρία Γιούσο. Έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς πολιτισμούς εδώ και αυτό έχει σημασία. Μιλάμε για ένα έθιμο αν θέλετε το οποίο περίπου ανήκει σε όλο τον κόσμο, χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο όπου υπάρχει το σταφύλι αλλά και όταν δεν υπάρχει το σταφύλι κάνουν μέσω ζυμώσεως προϊόντα είναι ο πνευματόδη από από διάφορα άλλα προϊόντα. Και φυσικά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι κατανάλωσης. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να αποφύγουμε εδώ να γελιοποιηθούμε γιατί ορισμένοι ε, προτείνουν πράγματα τα οποία είναι λίγο αστεία. Αν πιστεύουμε ότι με τις ετικέτες μπορούμε εμείς να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου, γελιοποιούμεθα. Όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Ντόρφμαν, όλες οι γυναίκες γνωρίζουν ότι όταν είναι έγκυες δεν πρέπει να πίνουν, δεν πρέπει να καπνίζουν και δεν πρέπει να πίνουν και καφέ, γιατί και η καφεΐνη όλοι οι γιατροί ε, λένε ότι δεν πρέπει να καταναλώνονται από εγγύους. Ε, οπότε τώρα τι θα βάζουμε πάνω στα κουτιά του καφέ ή στο ποτήρι, στην κούπα του καφέ. Ε, πραγματικά δεν υπάρχει καμία περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας όπου δεν παρακολουθείται τόσο στενά όσο κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου αυτής. Ε, γιατί υπάρχει τώρα πια μια, ένας έχουν δημιουργηθεί κάποιες συνθήκες φροντίδας της εγγύου με συνεχείς αναλύσεις, παρακολούθηση της δίαιτας και είναι γελίο το να πιστεύουμε εμείς ότι με τις ετικετούλες μας θα μπορέσουμε να δώσουμε οδηγίες ε, στα άτομα τα οποία βρίσκονται στην περίοδο της ζωής τους όπου είναι πιο στενά ελεγχόμενα από ότι ε, στην υπόλοιπη τους ζωή. Το πρόβλημα είναι οι εξαρτημένες γυναίκες από το ενόπνευμα οι οποίες δεν μπορούν να απαλλαγούν από την εξάρτησή τους αυτή και μόνο οι γιατροί μπορούν να τους βοηθήσουν. Δεν είναι θέμα ετικέτας. Το πρόβλημα λοιπόν και το λέγουν ε, οι ειδικοί, υπάρχει μια ένωση στην Ιταλία η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τις υπατικές ασθένειες και λέγουν ότι η βασική διαφορά στην εξάρτηση του ινοπνεύματος και στην κατάχρηση του ινοπνεύματος από τους νέους είναι οικογενειακής προέλευσης, πόσο παρακολουθούνται από τους γονείς τους τα παιδιά. Γιατί αν δεν παρακολουθούνται υπάρχει αύξηση κατανάλωτης 2-3% το πολύ όταν δεν ελέγχονται τα παιδιά από την οικογένεια, όταν δεν εκπαιδεύονται από την οικογένεια, τότε ε, νέοι ε, πραγματικά περνούν στην κατάχρηση με αυξήσεις κατανάλωσης πάνω από το 12%. Υπογραμμίζουν λοιπόν ότι το θέμα είναι θέμα εκπαίδευσης. Και το είδαμε εμείς ε, με τα δικά μας παιδιά που είναι οι πρώτες γενιές αν θέλετε των παιδιών που εφαρμόζουν όλους τους νέους κανόνες στη χώρα μου τουλάχιστον για την μη κατανάλωση πνεύματος ε, πριν από την οδήγηση. Στη χώρα μας επιτρέπεται μία μικρή δόση πνεύματος στο αίμα και αναφέρθηκε στα θέματα αυτά η Πιλάρα Ιούσου αλλά για τους νέους ε, κάτω των 21 απαγορεύεται πλήρως, όπως επίσης απαγορεύεται πλήρως και για τους επαγγελματίες οδηγούς, ε, μεταφορείς και τα λοιπά. Λοιπόν, τα παιδιά οργανώνονται, γνωρίζουν το πρόβλημα, όταν βγαίνουν το βράδυ υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν πίνει για να οδηγήσει ή οργανώνονται με τους γονείς τους για να τους γυρίσουν στο σπίτι το βράδυ. Υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν μέσα δηλαδή και ε, φυσικά όλα αυτά περνούν ως συνήθως από την εκπαίδευση. Το να βρει όλες αυτές τις οδηγίες σε μία ετικέτα αυτό θα καταστήσει γελία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε πραγματικά θα γυρίσουμε στα λεγόμενα τετράγωνα κολοκυθάκια. Κοιτάξτε, εμείς ε, ζητάμε πράγματα άχρηστα, ζητάμε πράγματα γελία. Δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί αυτό νομίζω θα σπρώξει πάρα πολλούς ε, Ευρωπαίου στον ευρωσκεπτικισμό. Ας είμαστε επιφυλακτικοί λοιπόν συνάδελφοι. Ας μην ξεχνάμε τι πολιτισμός βρίσκεται πίσω από ένα μπουκάλι κρασί. Την παράδοση της εινοπαραγωγής που συνδέεται με την ιστορία, την εινοπαραγωγή που συνδέεται με τη γεωπολιτική, με την μετανάστευση, με την ιστορία εν του λαού μας. Από τον ΝΟΕ είχαμε τα μπέλια. Λοιπόν, ας αποφύγουμε τη γελιοποίηση γιατί διατρέχουμε το κίνδυνο για μια ακόμη φορά να ενισχύσουμε αυτούς οι οποίοι είναι εναντίον της Ευρώπης. Ευχαριστώ Ελίζα Μπέτα. Φλόρενς. Ναι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όλα τα καλά επιχειρήματα που ακούστηκαν. Αλλά μόλις είχαμε ευρωεκλογέ και σε κάθε εκδήλωση, τουλάχιστον σε μένα, οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν ότι η Ευρώπη μπαίνει σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και θα με εξέπλητε ε, εάν ε, αυτό ήταν διαφορετικά στην Ιταλία ή στην Ελλάδα ή αλλού. Εμείς δηλαδή στις θα πρέπει να δώσουμε στην κυβέρνηση της ε, Γαλλίας συμβουλές ή στους Έλληνες πολίτες στην Αθήνα. Ε, ε, ξεσπάσουν σε γέλια. Ε, έχουμε κυβερνήσεις πάρα πολύ υπεύθυνες στις χώρες μας. Ας αφήσουμε να ε, το αναλάβουν αυτές και να μην ανακατευόμαστε εμείς. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φιλίπ Γου, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για να μας εκθέσει τις απόψεις της Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το ενδιαφέρον και η στήριξη του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της ΕΝΒΗ για τα θέματα που σχετίζονται με το ενόπνευμα είναι σημαντική για την Κομισιόν και καλοδεχούμενη. Η Επιτροπή έχει πλήρη συνέστηση ότι η κατανάλωση ενόπνευματος έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην υγεία και σε άτομα του περιβάλλοντος αυτών που δεν πίνουν η βία εντός των οικογένειων όπως υπόθηκε και γενικότερα στην κοινωνία. Η προσπάθεια από την ε, Ένωση, τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών είναι αναγκαίες. Αλλά παραπέρα, εφόσον πήρα το λόγο, να διορθώσω ορισμένες ε, ενδεχόμενες παρανοήσεις για το κείμενο που προτείνουμε. Στο σημείο 1 και 9 του ψηφίσματός σας, αναφέρεστε σε ένα πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το Ινόπνευμα. Ε, είναι σαν να έχουμε ε, εμείς ε, εγκρίνει πρόγραμμα για τη βλάβη που προκαλεί το ενόπνευμα. Εμείς ξεκινήσαμε κάποιες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κατανάλωση inoβλέματος από τους νέους και ιδιαίτερα πολύ έντονη σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εμείς ξεκινήσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του 2006 και οι προτάσεις μας ισχύουν. Κατά τη διαδικασία συζήτηση με τα κράτη-μέλη κατέστη σαφές ότι δεν μπορούσε το προηγούμενο σώμα των επιτρόπων να εγκρίνει κείμενο Είπαμε όμως ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε για ένα σχέδιο δράσης και ότι στοχεύουμε στα πλαίσια της στρατηγικής του 2006 να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Εγκρίναμε ένα διετές πρόγραμμα δράσης για τους ε, συνήθεις πότες και τους ε, περιστασιακούς πότες. Και είπαμε ότι θα στηρίξουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών βοηθώντας μαζί με τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την εφαρμογή αυτού του προγράμματος δράσης. Επιπλέον, και τα κράτη-μέλη επίσης θέλουν να σας ενημερώσω, εξετάζουν ποια θα μπορούσε να ήταν η ενωσιακή προοπτική και προσέγγιση. Και τον ε, προηγούμενο Δεκέμβρη ενέκρινε ένα κείμενο καθορισμού του πεδίου δράσης που εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες μας. Αλλά όπως υπόθηκε επανειλημμένα σήμερα εδώ. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι κύριοι υπεύθυνοι για το θέμα αυτό είναι τα κράτη-μέλη. Ο κανόνας μας ήταν και πάντα είναι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη όπου θα μπορούσε να υπάρχει ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Είμαστε τώρα στη φάση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω για τη βλάβη από κατανάλωση ενωπνεύματος Όλες προτάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους είναι καλοδεχούμενες και θα εκτιμηθούν στα πλαίσια της διαδικασίας που είναι εν εξελίξη. Τμήμα αυτής είναι πως η βλάβη αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί ολιστικά για να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα υγείας και να μειώσουμε τις επιπτώσεις των χρονίων νοσημάτων. Είναι προτεραιότητά μας αυτό. Μέχρι να διαμορφώσουμε την ε, πολιτική μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα με βάση την υπάρχουσα στρατηγική. Και θέλω να πω σαφώ γιατί ορισμένοι είπατε ότι έληξε το 12 η στρατηγική μα και γιατί δεν υποβάλλουμε νέε προτάσει, αλλά πολλά έχουμε κάνει έκτοτε. Συνεχίσαμε να διευκολύνουμε την εργασία και να επιτηρούμε τις διαδικασίες, την εργασία και τις διαδικασίες των κρατών μελών. Μέσω αυτής της Επιτροπής Εθνικών Αρχών και μέσω του Φόρουμ Ινόπνευμα ε, και Υγεία και στηρίζουμε και τα κράτη-μέλη στην εργασία που κάνουν για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα δράσης. Από πέρυσι συμβάλλουμε και σε κοινέ δράσεις για να μειωθεί η βλάβη από το ενόπνευμα. Τριετές που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα υγείας για να ανταποκριθούμε σε ορισμένα θέματα που θέσατε. Μπορούμε να συζητήσουμε για τους διαφορετικούς κανόνες από τα κράτη-μέλη μπορούν να υπάρξουν προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, ήδη σε διάφορα κράτη-μέλη, σήμερα ακόμη, είναι διαφορετικοί οι ορισμοί του κατοφλίου κατανάλωσης άνευ κινδύνου. Όλα αυτά συζητούνται μεταξύ κρατών μελών με τη στήριξη της Κομισιόν. Πρέπει επίσης ε, να εστιάσουμε εκεί που θέλουμε να έχουμε επίδραση. Υπάρχει μια διακυβέρνηση ομάδα του Φόρουμ η και Υγεία και να βελτιωθεί η λειτουργία αυτού του Φόρουμ. Καταλήγοντας, τονίζω, ότι η Κομισιόν συνέχισε με βάση τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές από το 2006 την εργασία για το θέμα αυτό και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας γιατί πρέπει να το αναφέρω και αυτό είναι σημαντικό. Και εξετάζουμε τη μελλοντική μας στρατηγική για το θέμα αυτό και ελπίζουμε στο ιδιαίτερα εγγύς μέλλον με βάση όλη την πληροφόρηση από όλους τους φορείς και από όλα τα κράτη-μέλη ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να διατυπώσουμε νέες προτάσεις και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 31 Μαρτίου και στην Ολομέλεια στη 2η του Απριλίου. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Το πρόγραμμα REFIT, πρόγραμμα ελέγχου καταλληλότητας και αποδοτικότητας της νομοθεσίας. Και να πάρω το λόγο εγώ ως εισηγητής τον, Μάιο, τον Ιούνιο του 2014 η Επιτροπή δημοσίευσε μία ανακοίνωση για το REFIT. Η κατάσταση και προοπτικές. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αποφάσισε μία έκθεση πρωτοβουλίας. Εμείς ε, θα γνωμοδοτήσουμε επ' αυτού. Το πρόγραμμα REFIT είναι μια εκθεση πρωτοβουλιας εμεις θα γνωμοδοτησουμε από αυτό. πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απλουστεύσει και να εξορθολογήσει το διακανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πρέπει να είναι ευκρινές, εύκολο στην κατανόησή του, να καταστέλει την γραφειοκρατία, να βελτιώνει την διατύπωση και την ποιότητα της νομοθεσίας έτσι ώστε να πετύχουμε τους στρατηγικούς στόχους που προσφέρονται από την οδηγία της Ένωσης στην χαμηλότερη δυνατή τιμή. Σεβόμενοι πλήρως τις συνθήκες και ιδιαίτερα σεβόμενοι τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία ελέγχου μέσω του REFIT που συνοδεύεται από την πρώτη έκδοση ενός ετήσιου δελτίου εποπτείας του REFIT που αναφέρεται στα ποσοστά εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Κάποιες από τις αρμοδιότητες είναι δικές μας, όπως η οδηγία για την ποιότητα του εδάφους και άλλες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, ο συνεχής έλεγχος για την προστασία των πτηνών στο Natura 2000, οι νέες αξιολογήσεις που έχουν ανακοινωθεί για, την, για, τον περιορισμό και την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα, η αξιολόγηση των χημικών ουσιών εκτός REACH. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σειρά ε, νομοθετικών πράξεων που έχουν πλέον θεωρηθεί απαρχαιωμένες. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να μειώσουμε την γραφειοκρατία, να μειώσουμε τα περινά γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά είναι θεμητή η ανησυχία μιας πλήρους απελευθέρωσης, ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος, της τροφιμικής ασφάλειας, και της υγείας γενικότερα. Σαν παράδειγμα, Εμφυμίστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αξιολογήσει την δυνατότητα να αποσύρει την οδηγία για τις πλαστικές σακούλες μετά τη συμφωνία των συνομοθετών επί της ουσίας. Όπως και η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για την αναθεώρηση ε, των κανονισμών για τα απόβλητα, όπως επίσης ε, και την μεταρρύθμιση ε, για τα συστήματα ελέγχου των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι ακριβώς λόγω αυτού του ιστορικού περιμένουμε από την, ενία, από την νέα επιτροπή, από τον αντιπρόεδρο Τίμερμαν στον Μάρτιο κάποια στοιχεία τα οποία θα μας διευκρινίσουν την κατάσταση. Είναι επίσης σαφές ότι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση που βρίσκεται υπό εξέταση θα βοηθήσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον συνάδελφο κύριο Καπούτο για τη σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την δουλειά την οποία έχετε ήδη κάνει. Το REFIT έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κατάργηση των διοικητικών βαρών της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα όμως δεν θα πρέπει να μειώνει τα ποσά που προορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας και γενικά αναφέρομαι στις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πλαστικές τσάντες και τα απόβλητα θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ορισμένα επιπλέον σημεία τα οποία θεωρώ κεφαλαιόδη και τα οποία οφείλω να υπογραμμίσω και θα καταθέσουμε τροπολογίες επ' αυτού. Καταρχάς το gold plating. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες ε, διευκρινίζουν περισσότερο τις προτάσεις ε, ε, οι οποίες γίνονται έτσι ώστε να δώσουμε πλήρη βεβαιότητα την ευρωπαϊκή παραγωγή μέσω ε, συγκριτικών ε, παρατηρήσεων. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δικαιολογήσουν την εισαγωγή αυτής της μεθόδου που δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Εφόσον θα πρέπει να προστατεύσουμε κάποια, σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο το περιβάλλον, απαιτούνται μελέτες και σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας δώσει περισσότερες εγγυήσει για την διαφάνεια σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων ε, μελέτης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και στις μικρομεσ... για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του δημοσίου στις διαβουλεύσεις, ε, πρέπει να είναι ελεύθερη η συμμετοχή και θα πρέπει να υπάρχουν και online επίσης ε, ε, διαβουλεύσεις. Τέλος, μεγαλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής μας, για να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση αυτών των συστημάτων απαιτούνται νέα μέσα όπως η διαδραστικότητα, τα open data ε, και τα cloud computing. Αυτό θα μειώσει και το κόστος σχετικά με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέσα και εργαλεία. Νομίζω ότι ακριβώς αυτές οι διαδραστικές χρήσεις θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκίρλινγκ. Ευχαριστώ για την εργασία που κάνετε για το θέμα αυτό. Η ομάδα μου τονίζει. ότι η διαδικασία αυτή είναι συνεχιζόμενη. Δεν είναι μόνο ένα θέμα που θα μας προσχολήσει μόνο μια φορά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ενταγμένο στην νομοθετική διαδικασία μια για πάντα. Οπότε θα θέλαμε κάποιο σχολιασμό ιδιαίτερα όσον αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων. Πιο πολλές λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ετήσιο κείμενο που να μας δίνει τη σχέση κόστους-οφέλους. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στον περιβαλλοντικό τομέα μια απλή διαδικασία για παράδειγμα όπως ε, η παραγωγή τυριού άμα δούμε πόσοι κανονισμοί εμπλέκονται που δεν αλληλοσυμπληρώνονται πολλές φορές ούτε καν συνδέονται λογικά και αν βάλουμε και κάτι για τα ζώα τότε γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο εκθετικά πιο περίπλοκο θέλουμε να αποφύγουμε να συνεχιστεί να υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι θα ήταν κακή για το περιβάλλον πιο απλή και πιο ευφυείς κανόνες. Θα ήθελα η Επιτροπή μας να τονίσει ότι θα είχε να ωφεληθεί το περιβάλλον από μια τέτοια απλούστευση. Διότι μέσω της απλούστευσης ε, μπορούμε να διασφαλίσουμε και καλύτερη συμμόρφωση. Και όπως έχουμε πει επανειλημμένα εδώ, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση, τι έννοια έχει να αποφασίζουμε μέτρα. Απλούστευση ίσον περισσότερη συμμόρφωση. Αυτός είναι ο στόχος οποιοδήποτε νομοθετήματος. Επίσης, μέσω της γνωμοδότησης να τονίσουμε πόσο σημαντικές είναι οι μικρομεσαίες. Αναφέρονται στην ανακοίνωση για το REFIT και σε άλλες γνωμοδοτήσεις επιτροπών, ζωτικότατες για τους ε, τομείς μας, παίζουν ε, ρόλο κλειδί για το λεγόμενο πρασίνισμα της οικονομίας, ιδιαίτερα της οικονομίας τροφίμων. Οι θετικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους είναι πολύ θετικές. Και το θέμα είναι ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ε, πάρα πολλούς ε, κανόνες και πώς συνδυάζονται από την ε, οπτική εκείνου που προσπαθεί να τις εφαρμόσει όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, συμφωνώ με αυτό που είπατε για τις πλαστικές σακούλες αλλά είναι προφανές ότι όλοι έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Η Επιτροπή μας έχει πολύ υψηλό ποσοστό νομοθετημάτων, νομοθετικής εργασίας και ξέρουμε πολλές φορές ότι η προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού δεν δίνει πάντα το σωστό αποτέλεσμα. Ορισμένε φορές, ε, τρεις ώρα το πρωί σε ένα τριμερή διάλογο, Μπορεί αυτό που αποφασίζεις για να επιτύχει συμβασμό να μην έχει πλέον καμία λογική. Άρα πρέπει να επανεξετάσουμε μέσω του Refit πολύ προσεκτικά την νομοθετική διαδικασία από αρχή μέχρι τέλους και όπου έχουμε νομοθεσία σε πολύ περίπλοκους τομείς και πολύ συχνά τα περιβαλλοντικά είναι περίπλοκα να προβλέψουμε ένα δεύτερο στάδιο της ε, νομοθεσίας δηλαδή να έχουμε μία μελέτη επιπτώσεων μετά την εφαρμογή και φυσικά όλοι μετά οι εμπλεκόμενοι ηλεκτρονικά όπως λέει ο κύριος Καπούτο να σχολιάσουν και μετά να δούμε τι θα γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειωθεί η ισχύ της νομοθεσίας αλλά θα είναι πιστεύω ευκολότερη εφαρμογή της. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Ουίτεμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ε, σας ως εισηγητή ε, για το έργο σας. Γενικά, ε, μας αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση αυτή για το Ρίφιτς και εκτιμούν και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Για μας φιλελεύθερους είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για μας είναι αυτό ουσιαστικότατο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και μόνο στη Γερμανία, 43% των εταιριών δηλώνουν ότι η ψηλή γραφειοκρατία είναι εμπόδιο για επενδύσεις και δημιουργεί και ανασφάλεια γενικότερα. Για να σας δώσω και κάποια παραδείγματα κοινοτικής νομοθεσίας. Το REACH είναι ε, μεγάλο άχθος και οικονομικό αλλά και γραφειοκρατικό ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες αλλά και το Natura 2000 σε περιοχές του Natura 2000 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία να αντιμετωπίσουν όσο και πολύ μεγάλη ανασφάλεια ε, για τις επενδύσεις και τα κοινωνικά ε, ζητήματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Γενικά υποστηρίζουμε το σχέδιο του εισηγητού και ε, καλωσορίζουμε την προσέγγιση, αλλά για την παράγραφο 3 έχουμε μια ερώτηση, όπως είπε και η κυρία Γκέρλινγκ, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει αποτελεσματική συγγνώμη, νομοθεσία που να αναγκάζει τα κράτη-μέλη και τις εταιρείε να συμμορφώνονται. Όταν έχουμε όμως επικαλύψεις και είναι διπλές ρυθμίσεις, ε, όταν ε, μία από τις δύο ρυθμίσεις έχει καταστεί ε, απαρχαιμένη θα πρέπει να καταργείται. Και τέλο, η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΡΙΦΙΤ αναφέρει τη δράση που αναβάνουν τα κράτη-μέλη, το λεγόμενο gold plating, που έρχονται με εθνική νομοθεσία να ε, επιβαρύνουν ε, την κοινοτική. Και το 1 τρίτο έχει διαπιστωθεί ε, της γραφειοκρατίας οφείλεται σε εθνικές ρυθμίσεις που έρχονται να επιβαρύνουν την ενωσιακή νομοθεσία. Όλα αυτά ε, είναι ε, άχρηστα και θα πρέπει να καταργηθούν για να είναι σωστός και ο πίνακας επιδόσεων του ρίφιτ. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρία Κονέσνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν για αυτό το θέμα και εσάς προσωπικά για τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι ουσιαστικά περιλαμβάνει όλα όσα συζητήσαμε τους τελευταίους μήνες. Το ρίφιτ είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικά νομοθετικά ζητήματα. Και ήταν πολύ χρήσιμο για μας. Εσείς ο ίδιος ήσασταν πάρα πολύ διπλωματικός στον τρόπο με τον οποίο συνοψίσατε ε, το θέμα και σας ευχαριστώ. Λίγα σχόλια έχω να κάνω. και το πρόγραμμα REFIT. Για να έχει νόημα αυτό, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και έχει νόημα να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτή η δυσπιστία ε, προκύπτει και από τις συχνές αλλαγές των νομοθετικών προτάσεων, των νομοθετικών πράξεων, έρχονται νέοι κανόνες ε, επί κανόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά θέλουμε να το αποτρέψουμε αυτό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως να γνωρίζει και τους κινδύνους ε, που μπορεί να ενέχει η απορρίθμιση, η κατάργηση ρυθμίσεων, δηλαδή ανετικές συνέπειες για παράδειγμα στο περιβάλλον. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και το... Ε, όταν το είδα στο κείμενό σας, ε, ομολογώ ότι κάπως τρόμαξα. Δεν θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα ως πρόφαση για να απορρίπτει ε, ε, νομοθετικές προτάσεις που δεν της αρέσουν. Δεν έχει ακόμα αναφερθεί αυτό, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, δηλώσει ότι το α ή το β ζήτημα Ε, είναι προβληματικό, αυτό μπορεί να εκφράζει απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμίε. Α πούμε, το δικαίωμα των πολιτών στο νερό. Ε, είναι μια πρωτοβουλία πολιτών την οποία θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαλεστεί το ρέφιτ για να ε, το αρνηθεί. Και είμαστε στη διαδικασία γνωμοδότηση αυτή τη στιγμή. Για μένα λοιπόν είναι απαράδεκτο να επικαλεστεί η Κομισιόν το REFIT για να απορρίψει μια τέτοια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, επειδή απλούστατα δεν είναι του γούστου της. Δεν έχουν πολλές ευκαιρίες οι πολίτες να επηρεάζουν την νομοθετική μας ε, διαδικασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι ούτε αυτό το ελάχιστο ε, δυνατότητα επιρροή των πολιτών δεν θέλει να το σεβαστεί. Αυτό για το συγκεκριμένο θέμα. Και ένα ακόμα ήθελα να προσθέσω. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται δεκτές κάποιες προτάσεις. Θα ήθελα να έχω κάποια ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δικές μας προτάσεις και τι συνέχεια δόθηκε. Γιατί σε κάποια κράτη-μέλη πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε την εξή κατάσταση. Πριν ακόμα τελειώσουμε την εφαρμογή, τη μεταφορά ενός νομοθετήματος, δρομολογούνται δύο και τρία για το ίδιο θέμα που περιμένουν να εφαρμοστούν. Και ε, όλοι ρίχνουν την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το νερό, και ε, το έδαφος, η σχετική νομοθεσία θα πρέπει ε, να μας απασχολήσει και να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες. Πολύ συχνά τα κράτη-μέλη έρχονται αντιμέτωπα με προσφυγές στο δικαστήριο επί παραβάση γιατί κάποιοι γραφειοκράτες έχουν πολύ περίεργο τρόπο ε, ερμηνείας των νομοθετημάτων μας. Το ξέρω ότι θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε ε, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά νομίζω ότι οι χώροι γραφειοκράτες προσθέτουν νέα εμπόδια. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν θα πρέπει οι γραφειοκράτε να αποφασίζουν για το πώ εμεί θα πρέπει να εφαρμόζουμε τη δική μας νομοθεσία. Ευχαριστώ. you know, chair, Θα είμαι σύντομο όπω πάντα, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω, λέω, να είμαι σύντομο. Αν και δεν θα σα εκπλήξω, ότι ενδιαφέρομαι πολύ. Όλοι συμφωνούμε ότι μία απαραίτητη γραφειοκρατία πρέπει να καταργείται. Όμως ε, μέσω του refit προσπαθούμε να καταργήσουμε τις ρυθμίσεις. Τελεία. Δεν έχει να κάνει με την κατάργηση αχρήστων διοικητικών βαρών. Είναι ένας νέος τρόπος να μειώνονται οι ρυθμίσεις. Γι' αυτό ε, η οργάνωση Business Europe και οι μεγάλες βιομηχανίες ε, προωθούν το θέμα αυτό. Οπότε, τους ακούω πολλούς να λένε για τις μικρομεσαίες, είναι το νέο κόλπο. Αν θέλετε να επιτύχετε κάτι, πρέπει να πείτε ότι θα βοηθήσει και τις μικρομεσαίες, γιατί όλοι αγαπούν τις μικρομεσαίες. να κάνω μια παράθεση από μια οργάνωση μικρομεσαίων. Αναφερόταν στην, ε, στο θεματολόγιο Στόιμπερ. Όταν τον περασμένο Σεπτέμβρη δημοσιεύθηκαν τα συμπεράσματα του Στόιμπερ, είπε ότι ακούγεται ωραία αλλά είναι καθαρά λαϊκισμός. Έτσι το βλέπουν οι μικρομεσαίες. Αυτό το θεματολόγιο είναι προσπάθεια των μεγάλων εταιριών. Αν θέλουμε να καταργήσουμε την άχρηστη γραφειοκρατία, να καταργήσουμε αυτήν και δεν προωθούμε κατάργηση του κανονιστικού πλαισίου. Και οι περισσότερες προσπάθειες που είδαμε τους τελευταίους μήνες είναι όλο και πιο πολύ προσπάθεια απορρίθμισης. Εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ένωση δίνει προστασία του περιβάλλοντος για τους πολίτες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω νομοθετημάτων. Και ναι, αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σε αυτούς τους νέους κανόνες. Περί αυτού πρόκειται. Εμείς το καλούμε αυτό προστασία του περιβάλλοντος. Άλλοι το λένε γραφειοκρατία και ενόχληση. Συγγνώμη, αλλά οι νομοθέτες αυτό πρέπει να κάνουν. Να μην πέσουμε λοιπόν στην παγίδα. Να μην δώσουμε εν λευκό εξοδότηση για την κατάργηση του κανονιστικού πλαισίου. Θα ήθελα να είναι περισσότερο αυτό στην ε, νομοδότηση, αλλά εμείς οι πράσινοι θα υποβάλουμε τροπολογίες που επαναλαμβάνω δεν είμαστε κατά της άχρηστης γραφειοκρατίας αλλά είμαστε κατά εν λευκό κατάργησης του ρυθμιστικού πλαισίου. Γιατί αναφέρεστε στις μικρομεσαίες. Θα διαπιστώσετε ότι ακόμη και οι μικρομεσαίες δεν θεωρούν ότι κάθε μέτρο είναι κακό. Και τώρα το γεγονός ότι ανατέθηκε στον κύριο Στόιμπερ να συνεχίσει την προσπάθειά του. Γιατί δεν έγινε καμία συζήτηση για το ότι τα προηγούμενα πορίσματα δεν υποστηρίχθηκαν από τέσσερις από τις 15 οργανώσεις που ε, υποτίθεται ότι έπρεπε να τη στηρίξουν. Και οι τέσσερις αυτές ήταν περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσει υγεία, οργανώσει καταναλωτών και συνδικάτα. Αυτές οι τέσσερις οργανώσεις δεν το στήριξαν. Άρα βλέπετε ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση αυτής της προσπάθειας. Πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε σωστά και να μην ε, την πατήσουμε ε, υποστηρίζοντας ε, τους στόχους ε, των μεγάλων εταιριών και όχι των μικρομεσαίων. Ο κύριος Λαφόντε. Αφρόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία ακούστηκαν για την αξιολόγηση του Ρεφίτ. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με αυτό. Έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα το οποίο θέτει στόχους ε, με τους οποίους ε, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Δεν πρέπει να υποβραδυνθεί η διαδικασία. Ελπίζουμε οι υποσχέσεις ε, να γίνουν σεβαστές και να συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις νομικές ρυθμίσεις οι οποίες παράγονται ιδιαίτερα και στη φάση της εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών στους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι δύσκολο λοιπόν να συμφωνήσει κανείς με τις γενικές αυτές απόψεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε και υπέρ ε, της προσπάθειας την οποία έκανε ο εισηγητής και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από τη μία αναγνωρίζουμε δηλαδή τη σημασία της διαδικασίας ε, αυτή καθεαυτή και από την άλλη σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις συνέπειες που μπορεί να προκληθούν στις ε, νομικές ρυθμίσεις που έχουν σχέση με την παραγωγή τροφίμων και με την υγεία. Όπως έλεγε και η κυρία Γκίρλινγκ θα συμφωνήσω μαζί της, απλουστεύω δεν σημαίνει ότι χειροτερεύω μια οδηγία. Ε, μπορεί μερικές φορές να συμβεί αυτό, αλλά όπως είπε και ο κύριος Έκχαουτ, το πρόβλημα, ο κίνδυνος είναι να περάσουμε σε μια πλήρη φιλελευθεροποίηση των νομικών ρυθμίσεων και αυτό είναι κάτι με το οποίο εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν υποστηρίζουμε τις γενικές προτάσεις τις οποίες κάνει η γνωμοδότηση αυτή και οι προτάσεις μας θα έχουν σαν στόχο να την πιο ισχυρή, πιο δεσμευτική σε αρκετά σημεία και θα τα πούμε μέσω των τροπολογιών μας, αλλά εκφράζουμε κυρίως την ανησυχία μας για την φιλελευθεροποίηση και ζητάμε να μην υπάρξει αυτή η φιλελευθεροποίηση. Καλές λοιπόν οι γενικές κατευθύνσεις αλλά ενίσχυση της, του περιεχομένου της πρότασης αυτής πρέπει να υπερασπιστούμε τις νομικές ρυθμίσεις και τις οδηγίες για το περιβάλλον, για την υγεία, για την ασφάλεια των τροφίμων ε, ταυτόχρονα αξιολογώντας ε, ε, μέσα στο χρόνο το πώς εφαρμόζονται. Ευχαριστώ κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομη. Βεβαίω και προφανώ υποστηρίζω το σχέδιο γνωμοδοτησή σα. Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι η Ευρώπη επικεντρώνεται στα ουσιώδη και δεν θέλει ε, μανιωδώς να ρυθμίζει τα πάντα. Θέλουμε αποτελεσματική νομοθεσία, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι χαλαρώνουμε τις προδιαγραφές ε, για την υγεία, το περιβάλλον και ό,τι έχει σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να παρακολουθείτε με το ποιο τρόπο εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία, διότι όταν εξετάζουμε διάφορες οδηγίες που ισχύουν βλέπουμε ότι μεταφέρονται με κακό τρόπο, με διαφορετικό ε, ανάλογα με τη χώρα, άρα έχουν και διαφορετικές επιπτώσεις. Και αυτές λοιπόν οι διαφορές δεν οδηγούν στην επιθυμητή εναρμόνιση, αλλά μάλλον σε προβλήματα ε, ανταγωνιστικότητας ε, στην οικονομία. Και προηγουμένως ε, μιλήσαμε για τις μικρομεσαίες, αλλά νομίζω ότι πέσαμε ε, σε κάποιες ε, στρεβλές καταστάσεις και κάποιος μίλησε για λόμπι. Εγώ είμαι από μια περιφέρεια που έχει πολλές μικρομεσαίες, δεν έχουν χρόνο να κάνουν λόμπι, αλλά μας επισημαίνουν ότι έχουν δυσκολίες να εφαρμόσουν κάποια νομοθεσία που πολλές φορές δυσκολεύονται και οι ίδιοι να καταλάβουν. Και είναι ευρωπαϊκή αυτή η νομοθεσία. Αν θα ήθελα κι εγώ να υπερβάλλω θα μπορούσα να μιλήσω για το υπερβολικό ε, λόμπι των μη κυβερνητικών οργανώσεων που μπορεί να έχουν καμιά φορά δίκιο αλλά άλλες φορές υπερβάλλουν. Θα ήθελα λοιπόν να ε, απευθυνθώ και να απευθύνω έκκληση στη σοφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πολλές φορές ε, το Κοινοβούλιο ζητά περιτέ και άχρηστε νομοθεσίε που οδηγεί αυτό σε ένα πληθωρισμό νομοθετικών κειμένων. Το είδαμε αυτό την περασμένη θητεία. Από την άλλη θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ προσιλωμένη στην ιδέα της κυκλικής οικονομία και περιμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα κάνει σχετική πρόταση που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη τα ερχόμενα χρόνια. Ευχαριστώ στο πολύ ο κύριος Γκρότε. Καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει καταντήσει σχεδόν θρησκεία. Ε, ε, ο, ο καθένας έρχεται εδώ και κατηγορεί τον άλλον και τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν φέρνουμε εμείς μια νομοθεσία, ένα κανονισμό, αυτός ο κανονισμός ε, ε καθιστά περί τους 28 εθνικούς νόμους. Δεν χρειάζεται λοιπόν ε, να ε, μας στιγωνόμαστε και να πέφτουμε ε, στα χέρια αυτών που κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι έρχεται από τις Βρυξέλλες είναι κακό και ότι κάνουμε εμείς είναι καλό. Και είναι κακό για να νομοθέτη να λύνονται όλα στο ΔΕΚ. Το βλέπουμε στο επενδυτικό πρόγραμμα τώρα του Ιούνκερ. Γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ, γιατί δεν έχουμε σχεδόν καθόλου έργα που να τελειώνουν το σχεδιασμό τους δεν χρειαζόμαστε ε, τε, ε, οργανισμούς, προγραμματισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Συμφωνώ με αυτό που πρότεινε ο κύριος Λαβία, αλλά δεν θα πρέπει καμιά φορά ε, να αυτομαστιγωνόμαστε για τη γραφειοκρατία. Γιατί οι δικοί μας τα Υπουργεία που κατηγορούν και καθιβρίζουν την ε, Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, πότε πήραν ένα τηλέφωνο την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Παράδειγμα, οι τοπικοί υπουργοί στα κρατήδια στη Γερμανία έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια νομοθεσία για τα παλιά ε, Στα Λούνα Πάρκ, ναι. Ε, ότι ε, θα πρέπει ε, όχι να καταργηθούν αλλά να επισκευάζονται. Και τώρα έχουν καταργήσει τα Λούνα Πάρκ σε πανηγύρια για σοπικές γιορτές και τα λοιπά και ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Θα πρέπει να οργανωθεί σωστά αυτό, αλλά καμιά φορά και εδώ απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σαν σάκος του box ή ε, όλοι ε, εκδικούνται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτονώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να δώσετε κι εσείς μια συνέντευξη τύπου και να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποιος ε, φταίει και τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να δείχνετε τέτοια συγκράτηση, να αντεπιθυνθείτε κι εσείς τα κράτη-μέλη γιατί την αξίζουν αυτή την επίθεση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Σχράια. Εγώ στο Κοινοβούλιο λιγότερες ε, ΜΚΟ ε, έχουν απευθυνθεί σε μένα και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, και τελικά περί τίνος πρόκειται. Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος. Πρόκειται για το περιβάλλον, πρόκειται για την υγεία και για διάφορες οδηγίες αλλά εθνικά ο καθένας δίνει το δικό του περιεχόμενο. Χαίρομαι πάρα πολύ με τη γνωμοδότησή σας, μπορούμε πολλά να κάνουμε. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Πρώτον, η οδηγία για τους σκοτόπους των πτηνών. Στην Ολλανδία εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ υψηλά είναι τα πρότυπα. Οι άλλες χώρες δεν το έχουν έκανε. Και στην Γερμανία φτιάχνουμε σύραγγες ενός εκατομμυρίου και ενάμιση και στη Γερμανία καταργούνται. και ε, ε, τα αντίστοιχα ισχύουν για διάφορες καλλιέργειες και ε, οποροκυπευτικά για το, το άζωτο. Το άζωτο ξέρετε είναι αέριο, δεν σταματάει στα σύνορα. Ε, ε, στη, τα αζωτούχα είναι μια πολύ σκληρή νομοθεσία στην Ολλανδία δεν φτιάχνουν πια στάβλους, ε, στη Γερμανία που είναι από την άλλη πλευρά ε, των συνόρων φτιάχνουν νέους ε, στάβλους και νέες εκτοφές. Ενεργειακό πιστοποιητικό χρειάζονται όλα τα σπίτια στην Ευρώπη, στην Ολλανδία αυτό γίνεται, σε άλλε χώρε όχι. Η αντίσταση στα αντιβιωτικά είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αμέσω μετά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ολλανδία ο ανέχο είναι σε επίπεδο ελαχίστων ποσοτήτων 0,0001, τα ίδια κάνουν και τα άλλα κράτη, στόχος μας ποιο είναι η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αλλά σε όλη την Ευρώπη να συνεννοούμαστε και να τηρούμε όλοι τις δεσμεύσει μας. Και όταν μια χώρα είναι πρωτοπόρος θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω μέχρι να την φτάσουν και οι υπόλοιπε. Και οι ε, κανονικοί άνθρωποι, οι πολίτες έχουν πολλή δουλειά ε, να κάνουν και εμεί για να του το εξηγήσουμε για να υπάρχει και να επανέλθει εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Περί όλων αυτών πρόκειται και σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να μας μιλήσει ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και παρακαλώ ε, να μην μακρηγορήσετε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Το REFIT δεν είναι προσπάθεια κατάργησης ε, του κανονιστικού πλαισίου. Οι στόχοι της πολιτικής μας παραμένουν θέλουμε να επιτύχουμε καλύτερα αυτούς τους στόχους, τους πολιτικούς που έχουμε καθορίσει. <coughs> Και να δούμε ποιο είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα των νομοθετημάτων μας. Όσον αφορά τις αποσύρσεις, το Κοινοβούλιο είπε να κάνουμε μία διαρθρωμένη διαβούλευση πριν υπάρξει απόσυρση, οποιαδήποτε. Και στο πρόγραμμα εργασιών μας του 2015 αναφέρουμε τις ενέργειες στα πλαίσια του refit που προβλέπουμε για φέτος. Όταν ε, ετοιμάζαμε το πρόγραμμα εργασιών μας, αναλύσαμε γύρω στις 450 προτάσεις και ε, συμφωνήσαμε επί 80 για απόσυρση ή τροποποίηση. Και είπαμε τότε ότι θα περιμέναμε να ακούσουμε την άποψη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πριν επισημοποιήσουμε αυτές τις αποσύρσεις. Και αυτή η διαδικασία είναι ένα εξελίξη. Και όταν ολοκληρωθεί θα ε, καταλήξουμε κι εμείς στην τελική θέση μας. Βεβαίως υπάρχουν ε, προβλήματα εφαρμογής και μεταγραφής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αναφέρθηκε αυτό το θέμα του gold plating, της επιχρήσωσης. Είναι θέματα που θα τα αντιμετωπίσουμε στην ε, αποτίμηση που κάνουμε ως Κομισιόν. Αλλά, να πω κάτι θετικό για το τέλος. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι ευφιέστερη και απλούστερη νομοθεσία ελπίζουμε να διευκολύνει την εφαρμογή της με τελικό στόχο τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ελπίζουμε επίσης ότι το REFIT θα είναι μια ευκαιρία για να Αφισβητήσουμε ορισμένες από αυτές τις παρανοήσεις ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι πολύ δαπανηρή για τις επιχειρήσεις. Αυτά θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια του Refit. Έτσι λοιπόν με θετικό πνεύμα σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την εργασία μας. Οπότε σας ευχαριστώ για την στήριξή σας. Προσβλέπω στην περαιτέρω εργασία και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους για τα ενδιαφέροντα σχόλιά τους. Να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες 5 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ 26 Μαρτίου, στην Τζούρι τον Ιούνιο και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Και τώρα το επόμενο θέμα, το οποίο είναι συνέχιση της εκδήλωσης I, της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για την νεολαία, για την νεότητα. Να παρακαλέσω τους προσκεκλημένους μας, Παλούμπο και Ζέγκ, να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Uh, Σύντομα θα πρέπει να σας υπενθυμίσω περί ποιες πρωτοβουλίας πρόκειται. Το ΆΙ οργανώθηκε τον προηγούμενο Μάιο για πρώτη φορά με τη συμμετοχή 6.000 νέων Ευρωπαίων που συζήτησαν τις ιδέες για μια καλύτερη Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνέχεια που δίδεται σε αυτό το συμβάν έχει σαν στόχο την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους προσκεκλημένους νεαρής ηλικία και τα μέλη. Ε, τις βασικές ιδέες θα τις παρουσιάσουν ε, οι φιλοξενούμενοι μας και θα συζητηθούν ε, τα εξής θέματα. Μηδενικά απόβλητα, καινοτόμες μέθοδοι, αλλαγή μορφής παραγωγής, ε, εκπαίδευση καταναλωτών και ευθύνες πολιτών. Θα υπάρξει μια σύντομη εισαγωγή αυτών των βασικών ιδεών από τους δύο νέους φιλοξενουμένους μας και στη συνέχεια θα υπάρξουν ορισμένα σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής. Θα δώσω αμέσως το λόγο για δύο λεπτά στον καθένα στους δύο φιλοξενουμένους. Και μετά θα κάνουμε τον πρώτο γύρο των σχολείων ερωτήσεων από πλευρά των μελών. Κύριος Παλούμπο. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Θα σας μιλήσω για το πώς θα δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Μία από τις προτεραιότητες ε, που είχαμε καθορίσει ήταν να μειωθούν τα τροφιμικά απόβλητα και η μεταφορά τροφίμων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό να δημιουργήσουμε βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό θα βοηθήσει και περιβαλλοντικούς στόχους, μείωση των εκπομπών διοξιδίου, λιγότερη συσκευασία, λιγότερα απόβλητα. Και είδα ότι έχετε και τη δική σας εκστρατεία για τα απόβλητα τροφίμων. Βλέπω ότι στην καφετέρια σας προσπαθείτε να το κάνετε αυτό. Τι μπορείτε να αξιοποιήσετε μέσω των προγραμμάτων για την κοινή γεωρική πολιτική και τα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου για βραχύτερε αλυσίδε εφοδιασμού και να ενθαρρύνεται συνεργασία μεταξύ γεωργών. Έτσι θα δημιουργήσετε και θέσει εργασία ε, σε διάφορε περιοχέ μέσω ίδρυση συνεταιρισμών για παράδειγμα. Ήδη συμβαίνει σε ορισμένε ε, περιπτώσεις, αλλά θα μπορούσε να συμβεί πολύ συχνότερα. Τι μπορούν να κάνουν τώρα οι ευρωβουλευτές για βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού, να ζητήσουν από την Κομισιόν να υπάρξει η ανακοίνωση για το βιώσιμο σύστημα τροφίμων, τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Αυτή ήταν μια προτεραιότητα που καθόρισαν. Είναι, είναι μια κοινωνία με μηδέν σπατάλη. Και θα ήθελαν επίσης να υπάρξει το πακέτο για την κυκλική οικονομία. Αυτό θα μείωνε και τα σκουπίδια από τρόφιμα. Θέλουμε λοιπόν μια κοινωνία με μηδέν σπατάλη, μηδέν απόβλητα, μηδέν σκουπίδια. Και πρέπει να συνεργαστείτε βέβαια και με τις άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Στέφαν Ζάνκ για, τις δεύτερες αδειές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλή ιδέα, αλλά έχει υψηλό συμβολισμό, υψηλή συμβολική αξία. Το συζητήσαμε πέρυσι στο I. Είναι ένας κανονισμός για να μειωθεί η χρήση χαρτιού και να χρησιμοποιείται μόνο ανακυκλωμένο χαρτί. Είναι υψηλή συμβολικής αξίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το σώμα εκπροσώπων των πολιτών. Άρα θα πρέπει να είναι υπόδειγμα για όλα τα άλλα θεσμικά όργανα και για την κοινωνία ευρύτερα. Αυτό λοιπόν προτείνει. Ζούμε σε ψηφιακή εποχή να μειωθεί η χρήση χαρτιού και να είναι μόνο εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να μιλήσουν τώρα τα μέλη. Ο Καρχάιν Φλόρενς. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε και τα είχα διαβάσει κιόλα. Πολύ σωστό πιστεύω είναι. Βεβαίως ε, πρέπει να μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα και η προστασία των πόρων διότι ευτυχώς η Ευρώπη είναι μεγάλης κλίμακας εξαγωγέας, εξαγωγέας μηχανημάτων, αυτοκινήτων κτλ. και πολλών άλλων. Αλλά βλέπουμε ότι παράλληλα πρέπει να εισαγάγουμε και ε, τεράστια ποσότητα πρώτων ε, υλών. Γιατί δεν έχουμε. Οπότε, επειδή δεν έχουμε πολλές πρώτες ύλες, μεταξύ των και τα χαλίκια. Οπότε η ανακύκλωση δεν πρέπει να είναι δευτερεύον θέμα. Πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας. Εγώ τώρα όλο και περισσότερο δεν χρησιμοποιώ χαρτιά. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν θα χρησιμοποιώ ποτέ, αλλά θα είμαι πολύ φιδωλός στην κατανάλωση χαρτιού. Και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο για τέτοια θέματα Είμαστε πολύ προσεκτικοί ακόμη και το νερό της βροχής το αξιοποιούμε. Δεν πάμε τόσο άσχημα, αλλά πολλά μπορούμε να κάνουμε ακόμη. Είμαι σίγουρος και αυτή η δική σας ε, πρόταση ότι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, να αυξηθεί η ευαισθησία μας για το τι πρέπει να επιτρέπεται. Πρέπει να μας ενδιαφέρει η χρήση λοιπόν των πρώτων υλών ηλελογισμένη. Τώρα κάτι το θλιβερό, ο κλάδος της ανακύκλωσης. Ο κύριος Ποτότσνικ είχε προτείνει ορισμένα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν πέρασαν. Κάνουμε κάθε προσπάθεια όμως εμείς στα πλαίσια της δημοκρατικής μας λειτουργίας τα θέματα αυτά να επανέλθουν και να μας υποβάλουν καλές προτάσεις. Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε σε αυτή τη συζήτηση ενδεχομένω μέσω του ίντερνετ και χαίρομαι που η νέα γενιά ασχολείται ακριβώς με αυτά τα θέματα για τα οποία και εμείς έχουμε εργαστεί νομίζω είναι ευκαιρία και για μας. Και κάτι ακόμη δεν είναι θέμα οποιασδήποτε πολιτικής κατεύθυνσης, είναι θέμα που μας αφορά όλους και πρέπει να μας απασχολήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ οι συνάδελφοι να σέβονται τον χρόνο που τους έχει δοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε μοιραστεί σε πολλές επιτροπές και χαίρομαι που ήρθατε εσείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το θέμα που θέσατε είναι πάρα πολύ ουσιώδες για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, αναφέρθηκε ο Καχάνης Φλόρεντ στο πρόβλημα που έχουν στην Ευρώπη της έλλειψης των πρώτων υλών. Ε, άλλα μέρη του κόσμου γίνονται πιο πλούσια και είναι καλό αυτό. Αναπτύσσεται μεσαία του τάξη, η οποία ε, αρχίζει να απολαμβάνει όσα απολαμβάναμε εμείς ε, εδώ και καιρό, αλλά ακριβώς επειδή φθήνουν οι πόροι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη σπατάλη. Αυτό αφορά τα πλαστικά μπουκάλια, το χαρτί και πάρα πολλά που μπορεί ο καθένας να κάνει και ατομικά αλλά και θεσμικά το κοινοβούλιο. Αλλά η κεντρική ιδέα θα πρέπει, θα πρέπει να είναι εξή. Επειδή στη φύση δεν υπάρχουν ε, απόβλητα, ε, θα πρέπει και στην κοινωνία να αποφεύγεται αυτό. Ε, η κυκλική οικονομία και η αντίστοιχη δέσμη είναι κάτι το οποίο περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα πράγματα ε, από πλευράς ε, σφαιρικής. Και το αρχικό αποτέλεσμα, ε, προϊόν μάλλον και το τελικό αποτέλεσμα, όλη η αλυσίδα παραγωγής και των γεωργικών προϊόντων, αλλά και πώς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας ως κοινωνία απέναντι στον πλανήτη. Και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αυτό να το έχουμε ως σημαία και έμβλημά μας. Δεν είναι μόνο οι περιβαλλοντικές ανάγκες, θα είπα και προηγουμένως, είναι και οικονομικό ε, αυτό το θέμα και οικονομική επιταγή μάλιστα. Και αν μπορούμε να συνδέσουμε τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία με την ε, υπεύθυνη χρήση των πόρων, πραγματικά θα έχουμε επιτύχει τον τετραγωνισμό του κύκλου. Και χαίρομαι που η νέα γενιά, η γενιά σας ε, ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα και ε, βεβαίως ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να τα προωθούμε και να συνέδεσουμε. Ευχαριστώ κυρία Μπέρντα. Ε, Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή περιβάλλοντο όταν σα είδαμε στο Στρασβούργο. Δεν είδατε πολλού βουλευτέ και είναι κρίμα αυτό πραγματικά. Και σα χαιρετώ και από το Κέντ ε, που είναι το πανεπιστήμιό σα και είναι στην ε, εκλογική μου περιφέρεια. Το ενδιαφέρον για την οικονομία και για την οικονομία χαρτιού βλέπετε ότι εδώ δεν χρησιμοποιούμε χαρτί. Έχουμε την ημέρηση διάταξη στο iPad, αλλά τι θα γίνει το iPad όταν ε, θα το αλλάξουμε. Και ξέρετε ότι δεν τα κρατάμε πολύ καιρό. Θέλουμε λοιπόν ένα δεύτερο πακέτο, γιατί το θέμα είναι πώς σχεδιάζεις. Έχουμε και αυτά εδώ τα μικρά ε, κουτάκια μεγάλα ε, τα δύο όμως και ενός ε, αποτελούνται από δύο υλικά που είναι ανακυκλώσιμα, πλαστικό και μέταλλο, καταλήγουν στα σκουπίδια. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τους χώρους αποθήκευσης απορριμμάτων, πρέπει να δούμε γενικά τον κύκλο ζωής των ε, υλικών και αυτό θα είναι δαπανηρό και για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές γιατί συμπεριλαμβάνουν ακριβώς το αρχικό κόστος. Όλα αυτά τα κάνουμε ούτως ώστε να δείτε πώς λειτουργεί η πολιτική. Και έχω μια ερώτηση λοιπόν. Θα είναι δύσκολη η εφαρμογή αυτών που συζητάμε και θα απαιτηθούν πολλά από όλους τους πολίτες. Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να έχουμε τη στήριξη του κοινού. Σε πέντε χρόνια όλοι πρέπει να επανέλθουμε ενώπιον των ψηφοφόρων για να τους πούμε, κοιτάξτε, αλλάξαμε τον τρόπο αγοράς και κατανάλωσης προϊόντων. Και αυτό θα σας βοηθήσει σε 20-30 χρόνια. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να περάσει αυτό το μήνυμα και όλοι μας πρέπει να δούμε πώς θα το ε, επιχειρήσουμε να το περάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ ένα λεπτό καθένας για να αντιδράσει. Οι κύριοι Μπίρτερ και ο κύριος Ντάνς αναφέρθηκαν στον κύκλο ζωής των προϊόντων. Πώς λοιπόν θα πείσουμε το κοινό τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Μα αυτός είναι ο δικός σας ρόλος των πολιτικών. Εσείς πρέπει να εξηγήσετε στους ψηφοφόρους σας τι κάνετε, τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά που γίνονται αργότερα. Χθε είδα ένα σκέτς για κάποιον που κάθεται μπροστά σε, μια, σε ένα τζάκι και λέει στα παιδιά κοιτάξτε είχαμε ένα πολύ ωραίο πλανήτη και δυστυχώς αυτό που θέλαμε να κάνουμε μετά ήταν απλώς να υπάρχουν κέρδη για τους ε, κεφαλαιοκράτες και άρα το θέμα είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Γιάνκε πώς θα πείσουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν. Αυτό θέλω να σχολιάσω. Οι οργανώσεις νέων ε, δεν αξιοποιούνται επαρκώς για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι αυτές οι οργανώσεις ε, δεν έχουν πολύ ψηλό επίπεδο πολιτικής συνειδητοποίησης αλλά γι' αυτό είναι τόσο όμορφες. Δεν έχουν ε, σκοπιμότητες είναι πολύ ιδεαλιστές και έχουν θαυμάσεις ιδέες. Για παράδειγμα, υπάρχει η γενιά του έρασμος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι επαρκής ο διάλογος που γίνεται με αυτήν την ε, γενιά. Οι πολιτικοί θα μπορούσαν να ασχοληθούν περισσότερο. Υπόθηκε ότι είστε νομοθέτες. Δεν είστε μόνο νομοθέτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στο κέντρο της προσοχής όλων των πολιτών. Άρα δεν είστε μόνο νομοθέτες, είστε σύμβολα της Ευρώπης. Άρα έχετε ευθύνη. Είπατε ότι ανακυκλώνετε το νερό. Α, δεν το γνώριζα. Αυτές τις ε, δράσεις σας πρέπει ε, να τις κάνετε γνωστές στους νέους και γενικότερα στην κοινή γνώμη. Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Και τώρα δεύτερος γύρος ιδεών να δώσω το λόγο στο Λεωνάρντο για να μας παρουσιάσει μια τρίτη ιδέα. Λοιπόν, η τρίτη ιδέα ήταν να επεκτείνουμε το χρόνο ζωής των προϊόντων. Μερικοί ευρωβουλευτές είπαν τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν οι νοοτροπίες αλλά υπάρχουν και δυνατότητες πολιτικής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα κίνητρα στις εταιρείες για να επεκταθεί ο κύκλος ζωής των προϊόντων. Για παράδειγμα να είναι η οικολογική, η πολιτική δημοσίου προμηθειών, του σχεδιασμού, αλλά και εγγυήσεις μπορείτε να δίνετε. Εγγυήσεις μπορούν να έχουν τα προϊόντα. Είναι σημαντική επίσης η κυκλική οικονομία, το συζητήσαμε, και αυτό μπορεί να βοηθήσει ως εργαλείο για να επεκταθεί ο κύκλος ζωής των προϊόντων, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες. Το βραβείο <clears throat> για την ε, κοινωνική καινοτομία θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα βραβείο για βιωσιμότητα, για προϊόντα με ε, μακρύτερο κύκλο ζωής. Το Κοινοβούλιο επίσης θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει πιλωτικά προγράμματα για τον προβλησμό του 16 Οπότε το κύριο κατά την επόμενη πενταετία είναι να προωθήσετε και να συμπεριλαμβάνετε στα νομοθετήματά σας τα θέματα του κύκλου ζωής, του μακρύτερου, της μακρύτερης διάρκειας ζωής των προϊόντων. Ξέρω ότι στη φάση του σχεδιασμού προκαλούνται πολλά στοιχεία περιβαλλοντικού κόστους, άρα να λαμβάνονται υπόψη και στο σχεδιασμό τα θέματα του περιβαλλοντικού κόστους αργότερα. Ευχαριστώ και ο Στέφαν για την τέταρτη ιδέα. Τέταρτη και τελευταία. Σύντομη και απλή. Μια εκστρατεία θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ενημερώσουμε τους μαθητές, τα σχολεία, για θέματα περιβάλλοντος, βιωσιμότητας. Γιατί το προτείνω αυτό. Μπορεί να φαίνεται προφανές. Όταν στα δεκαετία του 90 ήμουν μαθητής, τα θέματα του περιβάλλοντος ήταν τμήματα της, ε, των συνηθιών μας. Ό,τι κάναμε είναι «ζεις σε έναν πλανήτη, πρέπει να κάνεις, η συμπεριφορά σου να είναι βιώσιμη, μη σπαταλάς νερό. Αλλά οι νέοι τώρα το είδαμε στο ΆΙ <clears throat> δεν έχουν ε, πλέον αυτήν την οτροπία. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό προτείνω μια προσπάθεια. Κάποιος διάσημος για παράδειγμα να μιλήσει για τα θέματα αυτά του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας. Μια διασημότητα λοιπόν θα έχει υψηλή ορατότητα. Αλλά να απευθύνουμε και στην κοινωνία και στις ενώσεις ε, διδασκόντων, καθηγητών, γιατί πολλές από αυτές τις εκστρατείες ξεκινάνε και τελειώνουν στις Βρυξέλλες. Και είναι κρίμα. Οι οργανώσεις νέων έχουν κάθε καλή διάθεση αν υπάρξει ενημέρωση να την ε, μεταδώσουν θα ήταν πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ακούμε τους συναδέλφους τώρα. Ο κύριος Σλέκ πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αν μου επιτρέψετε θα συνεχίσω στα κροατικά. Γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι στην Κροατία που παρακολουθούν τη συζήτηση αυτή και θέλουν να δουν ποιο είναι το μήνυμά μας. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά βλέπω νέους ανθρώπους εδώ που έχουν προσκληθεί από το Κοινοβούλιο οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ της κυκλικής οικονομίας και της εκπαίδευσης για να γίνει η κυκλική οικονομία μία από τις προτεραιότητες της παρούσης κοινοβουλευτικής εντολής. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση ήδη από τον Υπιαγωγείο και να προχωρήσουμε στην προώθηση της ιδέας της κυκλικής οικονομίας. Έτσι θα βοηθήσουμε ε, τους ε, νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν προγράμματα καινοτόμα και είναι κάτι το οποίο επιθυμούν, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν εύκολα. Έτσι θα συνεχίσουν λοιπόν και την διαβίου κατάρτισή τους. Οι νέοι θα πρέπει να μάθουν πώς θα δημιουργούν προϊόντα τα οποία θα έχουν μακρύτερη διάρκεια ζωής Ε, όταν τελειώνει ένα προϊόν με μια συγκεκριμένη χρήση να υπάρχει και συνέχεια στη χρήση αυτή σε άλλου είδους ε, κατηγορίες προϊόντων. Έτσι θα διαχειριστούμε τους φυσικούς μας πόρους με πιο σωστό τρόπο. Τέτοιου είδους προγράμματα καινοτόμα θα είναι και ε, πιο ε, παραγωγικά, αποδοτικά σε επίπεδο ενέργειας και θα μειώσουμε και την κατανάλωση ενέργειας. Τέτοιου είδους μηνύματα λοιπόν θα πάρετε από πλευράς μας. Ε, μετακίνηση του πληθυσμού των νέων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωστή ενημέρωσή τους, καινοτομία, ακόμα και κυρίως στις χώρες οι οποίες δεν είναι στη φάση στην οποία βρίσκονται ήδη κάποιες άλλες. Έτσι θα ενημερώσουμε λοιπόν για την κυκλική οικονομία και θα διαμορφώσουμε ένα νέο πρότυπο, ένα νέο υπόδειγμα για τους νέους. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. θα ομιλήσω την Ιταλική. Κατανοώ το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκαν ε, οι νέοι προσκεκλημένοι μας για μια σωστή ενημέρωση και τη σημασία που έχει η σχεδίαση των προϊόντων. Εγώ ήμουν σχεδιάστρια και πράγματι μέχρι τώρα η παρουσίαση των προτάσεων μέχρι τώρα δεν ήταν απόλυτα ικανοποιητική. Όχι μόνο και σε σχέση με την ποσότητα των προϊόντων τα οποία καλούμεθα να χρησιμοποιήσουμε, αλλά ακόμα και με τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν οικολογική ε, χρήση. Πρέπει να υπάρξει μια νέα σχεδίαση της στρατηγικής μας της ε, κοινοποίηση των προτάσεών μας ε, γιατί οι κοινότητες θέλουν να είναι δημιουργικές ε, και θέλουν είναι πισμένες οι κοινότητες των πολιτών για την ανάγκη της καινοτομίας και των νέων πρακτικών, των χρηστών πρακτικών που έχουν σχέση με την παράταση της χρησιμότητας των προϊόντων, που έχουν σχέση με τη σωστή διατροφή, με την συγκατοίκηση ε, με τη συμμετοχή στα κοινοτικά πράγματα. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διάσταση η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την πολιτική και να της δοθούν περαιτέρω κίνητρα σε αυτήν την συμμετοχική αντίληψη. Ελπίζω λοιπόν ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά shared economy, η οικονομία της συμμετοχής. Κύριε Σκρότο, ευχαριστώ. Μου άρεσε στην τοποθέτησή σας αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Το κάνουμε και εμείς εδώ στην Επιτροπή. Ε, στο παρελθόν μετά από μια τέτοια συνεδρίαση είχαμε τρία τεράστια ε, κοντέινερ με χαρτί που πηγαίναν στα σκουπίδια. Ε, τώρα ε, το λύσαμε αυτό, φτιάξαμε ένα πόρταλ ηλεκτρονικό για να μπορεί ο κόσμος και όλοι οι συνάδελφοι να το βλέπουν. Δεν έχουμε κανένα χαρτί και είναι πολύ ε, μεγάλη πρόοδος. Δεν θα πρέπει όμως να επαναπαυόμαστε και να δούμε το επόμενο. Δηλαδή θα δούμε πόσο διοργανώνουμε εδώ τη δουλειά μας, το στόλο μας ας πούμε και πώς θα προχωρήσουμε. Και ε, ε, τα αυτοκίνητα φυσικά εννοώ. Ε, υπάρχει προγραμματισμένη ε, λήξη ε, της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος από τον κατασκευαστή. Ας πούμε στα συστήματα ε, κατά των καυσαερίων στο αυτοκίνητο. Μετά από 80.000 χιλιόμετρα κανονικά έλυγε η εγγύηση. 80.000 χιλιόμετρα ήταν εγγυημένο ότι θα ε, ε, ισχύει το εξάρτημα και μετά δεν υπάρχει εγγύηση. Εμείς το καταφέραμε αυτό να πάει από τα 80 σε 180.000 ή σε 150.000 χιλιόμετρα. Γιατί όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, αν μη τι άλλο, ελπίζεις ότι θα σου κρατήσει μέχρι τα 150-180.000. Αυτό μπορεί να κάνει η πολιτική. Να καταπολεμήσει την προγραμματισμένη λήξη ε, της ζωής ενός προϊόντος. Θα πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτό και ε, αυτή η ε, μηχανή παραγωγής ε, σκουπιδιών και κοπής χρήματος να σπάσει. Δεν δίνεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, αλλά εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σχέιερ, ευχαριστώ και χαίρομαι με αυτό που άκουσα. Αλλά έχω με τρία σχολεία συναντηθεί ήδη και πολλοί ε, εντύπωση μου κάνει ότι τα παιδιά δεν έχουν ιδέα για τα όσα κάνουμε εμείς. Εγώ κάθομαι εδώ, τους λέω και συνεδριάζω για το δικό σας μέλλον. Κάπου θα πρέπει να συναντηθούμε. Ωραία αυτά που λέμε για την αηφορία, για τη βιωσιμότητα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση στα σχολεία. Να ξέρουν οι μαθητές, εμείς τι συζητάμε. Είναι πολλοί οι παράγοντες, θα πρέπει ο καθένας να ενημερώνει τον άλλον, να ανταλλάσσουμε απόψεις και το πιο σημαντικό είναι Ε, να πω ότι ε, έχω δει ε, και πανεπιστήμια, έχω δει και μαθητές του γυμνασίου και μαθητές του δημοτικού. Λοιπόν, οι μαθητές του δημοτικού ηλικίας 7 έως 12 ήταν οι πιο συνειδητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Και τελευταία αντίδραση της κυρίας Κάντενμπαχ. Έχω ένα πρόβλημα γιατί μπήκα αργά και δεν άκουσα τις παρουσιάσεις σας. Αλλά χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, που είχαμε την δυνατότητα και προηγουμένως να σας δώσω στο Στρασβούργο. Οπότε, πολύ θα ήθελα να έρθει στο Ευρωπαϊκό τουλάχιστον ένας από εσά άλλη μια φορά το Σεπτέμβριο για παράδειγμα <clears throat> έχω δυνατότητα να σας καλέσω για τρεις μέρες. Πηγαίνετε παρακαλώ στην ιστοσελίδα μου να ξανασυζητήσουμε ως ένβη. Γιατί συνήθως το Σεπτέμβριο δεν σπουδάζετε; Όλα τα θέματα που θίξατε, <clears throat> ιδίω την προηγούμενη φορά, αποδεικνύουν ότι είστε πλήρως μέσα σε αυτόν τον αγώνα και νομίζω ότι εδώ εμείς στην ΕΜΒΗ, τουλάχιστον αυτοί που είμαστε παρόντες, εκτιμούν ιδιαίτερα την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ, λέει Και πάλι η Λεωνάρντο και Στέφαν. Ένα λεπτό ο καθένας. Σας ευχαριστώ. Θα αναφέρω δύο πρακτικές ε, για τις δυνατότητες παρέμβασης. Το 2016 μπορείτε να επανέλθετε αφού εφαρμόσετε αυτές τις απόψεις όταν συναντηθείτε με, τις, ε, με τους νέους και μπορείτε να αναφερθείτε στις νέες σας πολιτικές ή μπορείτε στις συναντήσεις σας με τα σχολεία. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι σε αυτές τις συναντήσεις αυτό που έκανε εντύπωση στις συζητήσεις ήταν η αηφορία και τι θα πρέπει να κάνουμε και όπως έλεγε ο κύριος Χρότε υπάρχει ένα θέμα με την παλαίωση των υλικών και έγιναν κάποιες μικρές ομάδες εργασίας και σε τοπικό επίπεδο οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα αυτά με επιμέρους λύσεις, κοινότητες ε, ε, συλλογικής διαχείρισης και χρήσης ε, και τα λοιπά. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον. Να πω επίσης ότι φέτος υπάρχουν πολλές δυνατότητες και με την αναθεώρηση για την Ευρώπη 2020 μετά το Μάρτιο και τις συζητήσεις τον Σεπτέμβριο ε, και την ε, αναθεώρηση της ΚΑΠ επίσης στο τέλος του χρόνου και γι' αυτό έχετε την δυνατότητα με αυτά τα θέματα και με αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, τη δυνατότητα να ενημερώσετε τις οργανώσεις των νέων στις εκλογικές σας περιφέρειες. Ακούω ότι υπάρχουν αρκετές πρακτικές θετικές πρόσκλησης ε, νέων στο Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά στο προηγούμενο ΆΗ 6.000 νέοι συναντήθηκαν και είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν τις ιδέες τους, να συζητήσουν με λίγους πολιτικούς ήταν λίγοι οι βουλευτές που ήταν παρόντες, σας ενθαρρύνουμε στην επόμενη συνάντηση να είστε εκεί, να μιλήσετε μαζί μας και να είμαστε σε επαφή. Πολλοί νέοι σήμερα είναι στρατευμένοι στον τομέα αυτό. Αν εμπλακείτε θα λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές των απόψεών σας και εγώ. Εγώ θα στείλω tweets και θα μεταφέρω αυτές τις απόψεις ε, σε πολλούς. Και η τελευταία παρατήρηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο, είναι ο τομέας της παιδείας. Ε, στην εκπαίδευση ε, θα πρέπει να συνεργαστείτε με τους εκπροσώπους των ε, εκπαιδευτικών στις πόλεις. Έτσι θα μπορέσουμε να ακούσουμε ιδέες για την σωστή παιδεία των νέων και στα πλαίσια της διαβίου κατάρτισης το ίδιο μπορεί να γίνει και για τις άλλες τις γενναίες. Σας ευχαριστώ που ακούσατε τις απόψεις μας. Ελπίζω να συναντηθούμε στην συνάντηση του επομένου έτους. Εγώ ευχαριστώ και τους δύο για την παρουσία σας, για την δυνατότητα που μας δίνετε να ακούσουμε τις ε, ιδέες σας και να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων <clears throat> με ταχεία ανταλλαγή επιχειρημάτων. Σαν πινκ πονγκ και θέλω να συζητήσω με τους συναδέλφους να έρχονται συχνά νέοι. Βέβαια, όχι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, <clears throat> κατά την οποία δεν είναι παρόντες περισσότεροι συνάδελφοι, αλλά σε άλλη φάση. <clears throat> Ευχαριστώ. Θα τα ξαπούμε σύντομα. πλαίσια διάταξη ανταλλαγή απόψεων με τον Μάρκ Σπρέγκερ που είναι διευθύνων ε, σύμβουλος του ECDC τον έχουμε καλέσει και θα μας δώσει μία επισκόπηση των δραστηριοτήτων ε, του οργανισμού του που δημιουργήθηκε το 2004 και που στόχο έχει να διαπιστώνει και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα υγείας που δημιουργούν οι <clears throat> λοιμώδεις ασθένειες. Όπως ξέρετε, φέτος είχαμε την κρίση του έμπολα και η δραστηριότητα του οργανισμού αυτού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ε, πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών είχε πολύ να κάνει με αυτήν την ε, επιδημία Θέλουμε λοιπόν να μας ενημερώσετε για με τι κυρίως ασχοληθήκατε ε, πέρυσι και ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις για του χρόνου. Παρακαλώ έχετε το λόγο για 10-15 λεπτά γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη χαρά είναι που είμαι παρόν εδώ και όντω ήταν μια χρονιά πολύ άξιο σημείο όχι μόνο γιατί έχει επανεκλεγεί και έχουμε νέο λοιπόν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή και έχουμε νέο επίτροπο λοιπόν, για την υγεία. Ήταν και η πρώτη χρονιά της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για τις μεταδόσιμες μεταδοτικές ασθένειες. Παρακαλώ τους συναδέλφους και τους νέους ε, αν θέλουν να συζητήσουν και να πάρουν φωτογραφίες να βγούνε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Παρακαλώ συνεχίστε. Ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο εισηγητής για αυτό το νέο νομοθέτημα είναι παρόν εδώ στην πρώτη σειρά και περιμέναμε και τα αποτελέσματα της πρώτης ανεξάρτητης αποτίμησης του οργανισμού μου. Και φυσικά είχαμε αυτήν την πρωτόγνωρη επιδημία έμπολα. Όπως είπε και ο πρόεδρος, για όσους ε, είστε νέα μέλη της Επιτροπής να σας παρουσιάσω τους τέσσερις κύριους στόχους της οργάνωσής μας. Πρώτα απ' όλα συλλέγουμε πληροφόρηση, επιτήρηση και επίσης ενημέρωση για τις επιδημίες, να έχουμε στοιχεία δηλαδή, να ξέρουμε. Δεύτερον, συντάσσουμε ταχείες ε, αποτιμήσεις κινδύνων και ε, επιστημονικές συμβουλές. Στηρίζουμε τα κράτη-μέλη για την ε, προετοιμασία τους και το τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό έχουμε ένα ανεπτυγμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για ε, την μικροβιολογία και την επιδημιολογία στον τόπο των επιδημιών. Να πω δύο λόγια για τη δημόσια υγεία πριν προχωρήσω. Γιατί είμαστε οργάνωση που ασχολείται με τη δημόσια υγεία. Αλλά η δημόσια υγεία μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ορολογιακό μηχανισμό που έχει πολλά στοιχεία, έχει πολλά ε, τμήματα, που, αλλά λειτουργεί μόνο εάν όλα αυτά λειτουργούν από κοινού. Για παράδειγμα, είδα ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την ε, κρίση έμπολα και είπατε ότι είναι σημαντικό σε αυτή τη γνωμοδότηση όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε, να θεραπεύσουμε την ασθένεια, αλλά να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα της διατροφής και εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Όταν ε, έγραφα την παρουσίασή μου, βεβαίως ε, στο κέντρο της προσοχής μας ήταν ε, το έμπολα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 22.500 ασθενείς και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο πραγματικός αριθμός. Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα και έχουν υπάρξει 9.000 θάνατοι ε, Γουινέα, 3.000 Λιβερία, 8.500 Σιέρα 10.000 και πάνω από 800 εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα ασθένησαν ήδη και πάνω από 500 απεβίωσαν. Σε μια χώρα όπως η Σιέρα Λεόνε υπάρχουν μόνο 8 χειρουργοί σε μια χώρα 6 εκατομμυρίων κατοίκων. Πολλοί εργαζόμενοι του υγειονομικού τομέα, υγειονομικό προσωπικό, δυστυχώς πέθανε. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως με την πολύ ε, υποβαθμισμένη υποδομή υγείας αλλά και με πολλές συνήθειες και επίσης με τους τρομερά καταστροφικούς εμφύλους πολεμού, Ποια είναι η βασική ανασχόληση του οργανισμού μας, να γίνει μια ταχεία αποτίμηση του κινδύνου της κατάστασης στην Αφρική και σε τι βαθμό θα μπορούσε να επηρεάσει την Ευρώπη. Το κάναμε αυτό. Αλλά στην ίδια τη Δυτική Αφρική πώς μπορούμε να αποφύγουμε, να προλάβουμε τα ξεσπάσματα τη ε, ασθένεια. Πρέπει να έχουμε σωστή στρατηγική που να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Να πάμε σε κάθε χωριό για να σταματήσουμε εκεί την επιδημία. Να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα ανείχνευση όλων των επαφών. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει καλό σύστημα υγειονομική περίθαλψη. Και δεν υπήρχε καθόλου καλό. Ωραία. Η ανταπόκριση τη ε, ε, ε παγκόσμια κοινότητα ε, υπήρξε μεν, αλλά δεν ήταν επαρκή και θα μπορούσε να υπάρχει και πολύ καλύτερη ε, διατομιακή προσέγγιση. Αλλά ούτε αυτό λειτουργήσε καλά. Άρα εξαιρετικές δυσχέρειες. Τώρα, να αναφερθώ επίσης στην επιστολή για τα καθήκοντα που έστειλε ο πρόεδρος Επιτροπής, ο πρόεδρος Επιτροπής στον Επίτροπο Αντρουκάητης. Η Επιτροπή βεβαίως ανέφερε δύο προτεραιότητες εκεί σε αυτήν την επιστολή. Βέβαια, πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε τις πανδημίες και να βοηθήσουμε τις δυνατότητες ε, ανταπόκρισης, αντίδρασης της Ένωσης. Παίζουμε κεντρικό ρόλο και για την ε, νομοθεσία 1082. Στηρίζουμε λοιπόν την Επιτροπή και τις υπηρεσίε της για τις δύο προτεραιότητες λοιπόν. Αλλά νέα, το νέο μας καθήκον ήταν να στηρίξουμε τον ε, νέο συντονιστή της Ένωσης για το έμπολα να αντιμετωπίσει την κατάσταση στις χώρες αυτές. Τώρα τι λέει η απόφαση 1082. Χορηγεί στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες δυνατότητε συντονισμού στην προπαρασκευή και, και την ε, συλλογή στοιχείων από τα κράτη-μέλη για να υπάρξει αυτή η προετοιμασία. Θα έπρεπε λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να μας δώσουν διαβεβαιώσεις ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένα. Ότι έχουν τα συστήματα για να αντιμετωπιστούν ε, τέτοια ξεσπάσματα διαμεθοριακής ε, ασθένεια καλά εργαστήρια. Έχουν ε, την κατάλληλη υποδομή για την διάγνωση. Έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να κάνει όλη την αλυσίδα επαφών των κρουσμάτων και έχουν τη δυνατότητα να απομονώσουν αποτελεσματικά και να θεραπεύσουν τα κρούσματα. Η οργάνωσή μου προσπαθεί να βοηθήσει την Επιτροπή που αποτιμά την πληροφόρηση που λαμβάνει από τα κράτη-μέλη. Βεβαίως εμείς δεν ελέγχουμε εάν και κατά πόσο είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη. Επίσης, Πάντα προσέχουμε αναδιόμενες μεταδοτικές ασθένειες όπως ε, η έμπολα. Το Δεκέμβριο του 2013 αρχίσαμε να ασχολούμεθα ιδιαίτερος με την ασθένεια αυτή. Ξέραμε ότι σε αγροτικές περιοχές, σε περιοχές υπαίθρου της ε, Γουινέας υπήρχαν κρούσματα μιας ε, άγνωστης μεταδοτικής ασθένειας. Και ήδη το Μάρτιο του 2014 επιβεβαιώθηκε πως ήταν έμπολα αυτό που έχουμε διαπιστώσει στη Γουινέα. Όσο αναπτυσσόταν ε, η ασθένεια, τόσο περισσότερο αυξάναμε τις δυνατότητές μας και τους πόρους που διαθέταμε. Και τον Αύγουστο φτάσαμε στο επίπεδο που μας επέτρεπε να αφιερώσουμε πόρους και προσωπικό. Είχαμε καθημερινές συναντήσεις τεχνικές. Είχαμε πάνω από 60 συνεδριάσεις της διαχειριστικής ομάδας υπό την ηγεσία μου για το θέμα αυτό. Και ήμασταν σε καθημερινή επαφή με την Κομισιόν, με τον ΠΟΗ και με άλλε οργανώσεις. Κατά το τελευταίο εξάμεινο, μεταξύ 40 και 60 εμπειρογνωμόνων μας εργάζονταν για το έμπολα καθημερινά. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Κάναμε πολλές ταχείες εκτιμήσεις κινδύνου, δώσαμε ε, επιδιομολογικές ενημερώσεις ε, και επίσης δώσαμε συμβουλές για το τι πρέπει να γίνει για αυτούς που πηγαίνουν στις χώρες αυτές, ε, πρέπει να υπάρχει έλεγχος για τους επιστρέφοντες, για αυτούς που ταξιδεύουν. Πήγα σε ένα πολύ καλά προετοιμασμένο, για παράδειγμα, νοσοκομείο στο Λουξεμβούργο. Με εντυπωσίασε. Είχαν πραγματικά κάνει όλα όσα έπρεπε. Με ρώτησαν, κοιτάξτε, έχουμε όλες διαδικασίες ακριβώς εκεί. Αλλά εάν έχουμε ένα ασθενή, κάθε μέρα θα έχουμε πολλά απορρίμματα. Για παράδειγμα, όλες τις στολές που θα έχουν χρησιμοποιηθεί. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα απόβλητα. Απλή ερώτηση, αλλά δύσκολη απάντηση. Άλλη ερώτηση. Έχουμε πολλά, πολλά καλά συστήματα ιατρικής διακομιδής. Αλλά τι θα γίνει μετά, όταν ε, φτάσει ο ασθενής, μετά πώς θα γίνει η του αεροσκάφους. Και αυτό είναι περίπλοκο. Έχουμε δώσει πολλές τεχνικές συμβουλές, τις οποίες στείλαμε και στην Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας. Πρέπει να πω λοιπόν ότι η Επιτροπή αυτή και ο κανονισμό 1082 έπαιξε ουσιώδη ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Επίσης στείλαμε προσωπικό στη Δυτική Αφρική. Όχι τόσο πολλού. γιατί είναι σημαντικό να έχεις ε, από πρώτο χέρι πληροφόρηση. Τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο πρέπει να πω όμως ότι αυξήθηκε τόσο πολύ η πίεση να κάνουμε περισσότερα στη Δυτική Αφρική για να αλλάξει ισοδός κατάσταση. Και υπήρξε ένα ειδικό αίτημα του ΠΟΗ και από την οργάνωση στην Απλάντα ότι χρειάζονταν ε, γαλόφωνο προσωπικό. Εμείς έχουμε πολύ, πολλούς γαλόφωνους. Και οι δύο επίτροποι επίσης ε, σε εκείνη τη φάση επισκέφθηκαν τη Δυτική Αφρική και είδαν με τα μάτια τους ποιες ήταν οι ανάγκες επιτόπου. Κατόπιν λοιπόν ο Επίτροπο Ανδρουκάητης ήρθε στο, στα γραφεία μας αρχές Δεκεμβρίου και μας ρώτησε μπορείτε να εκπονήσετε ένα σχέδιο πώ να στηρίξουμε τη Δυτική Αφρική ιδιαίτερα στη Γουινέα που χρειάζονται γαλλόφωνου. Οπότε επειδή ήδη προετοιμάζαμε ένα πρόγραμμα πολύ σύντομα το είχαμε έτοιμο. Και ο υπεύθυνο για τις ε, λοιμώδεις ασθένειες, ο κύριος Κολομπιέ πήγε με άλλους εμπειρογνώμονες στη Δυτική Αφρική για να εφαρμόσει το σχέδιο αυτό. Και στα μέσα Δεκεμβρίου υποβάλαμε ένα σχέδιο στην Επιτροπή που προέβλεπε ότι θα έπρεπε να έχουμε τέσσερις ομάδες πεπειραμένων ε, εμπειρογνωμόνων και νέων εμπειρογνωμόνων που θα πρέπει να πάνε στις διάφορες περιοχές της Γουινέας για να στηρίξουν ε, τις τοπικές αρχές. Όχι για να περιθάλψουν, αλλά για να πάνε σε κάθε χωριό για να δουν ότι η βασική επιδημιολογική δουλειά γίνεται με τον σωστό τρόπο. Σήμερα έχουμε ήδη πάνω από τέσσερις ομάδες στη Δυτική Αφρική και χαίρομαι που και άλλες ε, χώρες ευρωπαϊκές έχουν στείλει προσωπικό στη Γουινέα για να αλλάξουμε την κατάσταση. Τώρα, πώς θα έχουμε πάει. Η νομοθεσία για διαμεθοριακά θέματα υγείας μας βοήθησε πολύ. Συνεργαστήκαμε τα κράτη-μέλη για το επίπεδο προετοιμασίας τους και νομίζω ότι και η Επιτροπή για την Ασφάλεια Υγείας έπαιξε ουσιώδη ρόλο για το συντονισμό τη διαχείριση του κινδύνου. Και επίσης οι κοινέ προμήθειες υλικού είναι πολύ σημαντικές. Θα έλεγα ότι δώσαμε όλα όσα χρειάζονταν. Επιτήρηση, στήριξη της προπαρασκευής, κατάρτιση, ενημέρωση και επαφές ε, μεταξύ πολλών χωρών και εδώ πολύ καλά τα πήγαμε, είχαμε πολύ χρήσιμες επαφές οι οποίες δεξίχθησαν με πολύ συντονισμένο τρόπο. Τώρα τα καθήκοντα του Επιτρόπου. Ήδη αναφέρθηκα σε αυτό. Στην ακρόαση που έγινε εδώ με τον Επίτροπο Αντρουκάητης είπε ότι πρέπει να προωθήσουμε, να προστατεύσουμε και να προλάβουμε. Θαυμάσιες πρωτοβουλίες αυτές. Αυτά είναι πολύ χαρμόσυνα για κάποιον όπως εγώ. Είμαστε κέντρο και πρόληψης και ελέγχου όπως είπα. Και θέλω λοιπόν να αποτύσω ιδιαίτερο φοροτιμή στην Ιταλική Προεδρία που έθεσε πολλά θέματα λιμουδών ασθενειών στην ημερήσια διάταξη. Είχαμε πολύ καλές ε, συναντήσεις για την υγεία στη Μεσόγειο, για το HIV και άλλα. Και υποστηρίζουμε και την Λετωνική Προεδρία που προσπαθεί να κατοπολεμήσει τη φυματίωση στην Ευρώπη. Και φυσικά θέλουμε να σας στηρίξουμε γιατί ξέρω ότι ασχολείται με την ε, ασφάλεια των ασθενών και τις αντιστάσεις στα αντιβιωτικά. Όταν ανέλαβα πριν από πέντε χρόνια η πρώτη μου προτεραιότητα ήταν να βοηθήσω να δημιουργηθεί ένας οργανισμός της που να είναι αξιόπιστος, που να θεωρείται χρήσιμος από τους πολίτες της Ευρώπης. Και χαίρομαι που ένα από τα πορίσματα τη εξωτερική ε, αποτίμηση είναι ότι τα προϊόντα μας είναι καλή επαγγελματικής ποιότητας σε όλους τους τομείς της εργασίας του. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι αν δεν είμαστε αξιόπιστοι, αν δεν ακούγεται η φωνή μας ε, με σοβαρότητα, δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε κανένα ρόλο γιατί δεν έχουμε επίσημε αρμοδιότητε. Χαίρομαι πολύ που η Διοικητική Επιτροπή μα εκπονεί τώρα συστάσει, διότι ω οργανισμό πρέπει να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές από τη διαχειριστική μας επιτροπή για την μικροβιολογία για την τεχνολογία πρώτης γραμμής και για τις μικρές χώρες και βεβαίως και οι δραστηριότητες ενημέρωσής μας το θέμα διαρροής εγκεφάλων και οι ανισότητες στα προγράμματα κατάρτισης. Τώρα στο μέλλον υπάρχουν τουλάχιστον 7 απειλέ που πρέπει να μα απασχολήσει. Η πρώτη είναι η αντίσταση στα αντιβιωτικά, δεύτερη είναι οι επιδημίες που προκαλούνται από διαβιβαστές, δεύτερον η αντίσταση στα εμβόλια και η φυματίωση. Η Ευρώπη έχει τεράστια πολυμορφία Πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να λάβουμε υπόψη επίση ότι θα συνεχιστεί η οικονομική αβεβαιότητα σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Καταλήγοντα, η οργάνωσή μα θα υποστηρίξει την νέα επιτροπή και τον νέο επίτροπο στα καθήκοντά του. Ο δόκτωρ Άντριου Κάιδη μα επισκέφθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Στοκόλμη και τον διαβεβαίωσα προσωπικά γι' αυτό. Δεύτερον, η νομοθεσία για τι σοβαρέ διαμεθοριακέ απειλέ υγεία που εσεί συνδιαμορφώσατε δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ισχυρό πλαίσιο για συνεργασία και συντονισμό. Θεωρούμε ότι η κρίση έμπολα επιβεβαίωσε την αξία αυτού του νομοθετήματο Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και να σα συγχαρώ για την προνοητικότητά σα. Η στήριξη τη Κομισιόν στην εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία είναι φυσικά η πρώτη προτεραιότητά μα. Τρίτον, Φέτος ε, είναι η δέκατη επέτειος της ε, δημιουργίας μας. Για δέκα χρόνια παρακολουθούμε, αποτιμούμε και ενημερώνουμε για τις λοιμώδεις ασθένειες, τους κινδύνους λοιμωδών ασθενειών στην Ένωση και τα κράτη-μέλη. Για τα επόμενα δέκα χρόνια η οργάνωσή μας θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για απρόβλεπτους κινδύνους και να βοηθάει τα κράτη-μέλη της Ένωσης στην προετοιμασία τους. Κλείνω αυτή την σύντομη παρουσίαση με μία μεταφορά. Είμαι Ολλανδός στη χώρα μου. Το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας είναι υπό το επίπεδο της θάλασσας. Αν υπάρχουν λοιπόν ισχυρές ε, καταιγίδες φοβόμαστε για τα φράγματά μας. Γιατί αν σπάσει ένας και, ένα και μόνο φράγμα θα έχουμε τρομερές πλημμύρες. Στον τομέα των ε, λιμωδών ασθενειών η Ευρώπη έζησε πολλές καταιγίδε τα τελευταία χρόνια. Το έμπολα ήταν μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη καταιγίδα. Αλλά κάθε φορά οι άμυνες της Ένωσης, τα συστήματα δημόσιας υγείας, άντεξαν. Είναι όμως αρκετά ισχυρά για να αντέξουν ε, την επόμενη θύελα ή τη μεθεπόμενη. Στην Ολλανδία ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να προσέχεις το πιο αδύναμο σημείο, το πιο αδύνατο φράγματος γιατί όλη μας η άμυνα είναι τόσο ισχυρή όσο το πιο αδύναμο συμμετή. Τον Νοέμβριο παρακολούθησα τη συζήτησή σας για το έμπολα. Συμφωνώ απόλυτα ότι η εστίαση της καταπολέμησης του έμπολα πρέπει να είναι στη Δυτική Αφρική και εργαστήκαμε με βάση τα πορίσματά σας. Πιστεύω λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος να υπερασπιστούμε τους πολίτες της Ένωσης από τις λοιμώδεις ασθένειες είναι να στηρίξουμε την πρόληψη και τον έλεγχο στην Ένωση και ευρύτερα και να παίξουμε, να ε, δώσουμε ειδική προσοχή στα πιο αδύνατα σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κονέτσκα. που είναι για την Επιτροπή μας το πρόσωπο που έχει την επαφή με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σπέγγλερ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα είμαι ιδιαίτερο σύντομη. Νομίζω ότι ο κύριος Σπέγγλερ ε, είπε αυτά τα οποία ε, έπρεπε να πει, δηλαδή εννοώ ότι είχε ουσία για τις εργασίες ε, της υπηρεσίας του. Η υπηρεσία αυτή δεν παρακολουθεί απλά, δεν εποπτεύει απλά, αλλά κυρίως προσπαθεί να βοηθήσει. Αυτός είναι ο στόχος του και αυτό κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπάρχουν νέες απειλές οι οποίες έχουν έρθει στην επιφάνεια και νέες προκλήσεις για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχου. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους πόρους τους οποίους διαθέτουμε στην συγκεκριμένη υπηρεσία και αν είναι δυνατόν να διευρύνουμε και τις αρμοδιότητές της. Εδώ υπάρχει ίσως κάτι περισσότερο συγκεκριμένο, το οποίο έχω πει στο παρελθόν, το Νοέμβριο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε ότι ο ρόλος του ECDC είναι ένα σημαντικός ρόλος και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες σε χώρες όπως η Μολδαβία, η Γεωργία, η Ουκρανία, γιατί όχι, οι χώρες οι οποίες σε κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οποίες δεν βοηθάμε όσο θα έπρεπε. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τις λειτουργίες, ε, τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου οργάνου και σε αυτές τις χώρες, οι οποίες πολλές φορές είναι ανίκανες καν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μαζί μας. Ένα άλλο σημείο το οποίο νομίζω ε, ενδιαφέρει όλους. Σήμερα ψηφίσαμε την απαλλαγή για το δημοσιονομικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά εμφανίζονται νέες απειλές. Τα χρήματα όμως τα οποία παίρνει η υπηρεσία δεν αυξάνονται. Είναι καλό κάποιες υπηρεσίες να έχουν την έδρα τους σε άλλες περιοχές όπως η Σουηδία αλλά αυτό είναι μερικές φορές ένα πρόβλημα. Ε, γιατί σε δημοσιονομικό επίπεδο αυτό αποτελεί ε, μια επιβάρυνση την οποία δεν αντιμετωπίζουμε εύκολα. και όλα γίνονται και με τις, ε, γνωρίζετε ότι χρησιμοποιείται άλλο νόμισμα στη Σουηδία Πολλές φορές ε, η αλλαγή των νομισμάτων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην ε, υπηρεσία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτά τα θέματα ακούγονται ίσονος σημασίας, αλλά παρόλα αυτά είναι θέματα τα οποία καλούμε θα αναλύσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Θα κλείσω λέγοντας ότι η Διαχειριστική Επιτροπή της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνει και δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα επιλέξει ένα νέο διευθυντή τον Μάρτιο αυτού του έτους για να αναλάβει τα ενία της συγκεκριμένης υπηρεσίας και νομίζω ότι ε, και εμείς θα μπορέσουμε να πάρουμε μέρος στην επιλογή και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να είμαστε παρόντες στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια εγώ θα ενημερώσω την Επιτροπή μας έτσι ώστε όλοι να έχετε στη διάθεσή σας τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε. είναι μία από τις μικρότερες εξωτερικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί ε, είναι μια υπηρεσία η οποία έχει βρει τη σωστή της θέση στην διοικητική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαιτέρως μετά από το ξέσπασμα της επιδημίας ε, ε, του ιού εμπόλα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε την επαϊοσύνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και Σπέγκλερ για την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ε, θέλω επίσης να ευχαριστήσω και όλα τα άλλα μέλη ε, της υπηρεσίας σας και νομίζω ότι μπορώ το ευχαριστώ αυτό να το πω από τα μέλη της, από πλευρά των μελών ε, του συνόλου της Επιτροπής μας. Να ευχαριστήσω αυτούς τους συγκεκριμένους συναδέλφους οι οποίοι έχουν μείνει μέχρι τέλους και ακούνε ε, τη συζήτηση αυτή. Επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση αυτή αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι μια σημαντική εξωτερική υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γκρότε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπρέγγερ, για την παρουσίασή σας. Ακούγοντας όλα αυτά, θα πίστευε κανείς ότι ε, έχει εκριζωθεί τελείως η έμπολα και η Ευρώπη έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς έλειπαν και τα στοιχειοδέστερα. Ήταν απόλυτη αποτυχία αυτό που ζήσαμε στην Αφρική. Ούτε γάντια δεν είχανε, ούτε τα στοιχειώδη δεν είχαν οι άνθρωποι. Και μάλιστα να μας προβάλλεται τόσο ρόδινα, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε στο μέλλον πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις. Γιατί σε αυτή την κρίση δεν αντιδράσαμε καλά και σωστά. Και ενδεχομένως ο οργανισμός σας να συνεισφέρει και προς την κατεύθυνση αυτή για το πώς να αναγκάσουμε στο μέλλον να μην υπάρξουν τέτοιες καταστροφές και τέτοιες όλες. Για να βάλουμε και λίγο νερό στο κρασί μας. Δεν τα πήγαμε καλά. Είναι σαφέστατο αυτό. Το συζητήσαμε και στην Επιτροπή μας αυτό. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά δεν μου άρεσε ε, ο τρόπος που ε, αντιδράσαμε. Ίσως να μας γίνει το, το πάθημα μάθημα. Για το μέλλον τώρα. Έχετε ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα εργασιών πώς διαμορφώνεται. Τι συντονισμός υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι γίνεται με τους άλλους οργανισμούς. Υπάρχει γιατί και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων ασχολούνται και με τον έμπολα και υπάρχουν κάποια σημεία όπου οι δύο προσπάθειες τέμνονται. Ε, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μας ενημερώνατε πώς συντονίζεστε και πώς διαμορφώνετε το πρόγραμμα εργασίας σας. Μόνοι σας συντονίζεστε με κανέναν, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με άλλους οργανισμούς ευρωπαϊκούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σχρέα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Σπρέγκερ ε, για την κατάσταση ε, και πώς την αντιμετώπισε. Και τον Νοέμβριο ήμουν παρούσα στη συζήτηση και ρώτησα τι γίνεται. Συμφωνώ απολύτως ε, με την πρώτη εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου. Ε, εντάξει, θα πρέπει να συνεχίσουμε μαζί στη συνεργασία, δεν μπορώ να τα επαναλάβω όλα. Ε, ε, συμφωνώ και με τον κύριο Γκρότε ότι χωράει βελτίωση, μα γι' αυτό βρισκόμαστε εμεί εδώ και το συζητούμε και θα πρέπει να το εντοπίζουμε. Και πώ θα μπορούσατε ε, να έχετε καλύτερη συνεργασία με το Γραφείο Ανθρωπιστική Βοήθεια. Έχω. Η φυματίωση επελάβνη, το ξέρετε, το έχετε υπόψη σας. Να μην έρθουμε του χρόνου να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα και η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και στην Ευρώπη αυτό και στην Αμερική. Κοιτάξτε τι λέει ο Ομπάμα στο θέμα αυτό της αντίστασης στα αντιβιωτικά ε, έχει να κάνει και με την υγεία ε, των ζώων ε, και τα τρόφιμα αλλά και για των ανθρώπων έχει σημασία. Εκεί υπάρχει κανένα συντονισμός. Μπορείτε εσείς να επέμβετε για να επηρεάσετε τις καταστάσεις. Ο κύριος Παρνιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά. Σε ό,τι με αφορά εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων σε αυτή τη πολύ σοβαρή και βαριά περίπτωση του έμπολα αντέδρασε και με την Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας και με τον οργανισμό σας. Έχουμε συνεργαστεί. Είναι στο Λουξεμβούργο η Επιτροπή και εμείς μάλιστα την ιδρύσαμε. Εγώ ήμουν και εισηγητής για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές για τη δημοσιακή και τώρα πριν από ένα χρόνο περίπου εγκρίναμε αυτή μας την απόφαση και ενισχύσαμε το συντονισμό που είναι και απαραίτητος μεταξύ των κρατών μελών και ε, του δικού σας οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα σε αυτό ε, το νέο όργανο, την Επιτροπή και θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μόνιμες και διαρκείς επαφές όταν ήμουν εγώ εισηγητή, συνεργάστηκα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και νομίζω ότι με τη νέα αυτή επιτροπή και τη δική σας δουλειά ε, έχουμε φτιάξει ένα ανάχωμα πολύ καλά κατασκευασμένο. Αλλά όπως το είπατε και εσείς ο ίδιος, θα πρέπει να προσέχουμε ε, τον ασθενέστερο κρίκο μια αλυσίδα. Και πραγματικά υπάρχουν πολλοί ασθενείς κρίκοι ιδιαίτερα στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Η Γενική Διευθύντρια στις 25 Ιανουαρίου τελικά αναγνώρισε ότι καθυστέρησε να καταλάβει πόσο σοβαρή ήταν η επιθυμία και ε, αυτή η επιθυμία και ε, οι ελλείψεις πρέπει να ε, τις γίνουν μάθημα. Τέσσερις ήταν οι ελλείψεις, οι ολιγορίες που επηρέασαν σοβαρά και τη δουλειά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτή τη μάστιγα που είναι ο ιός έμπολα. Γι' αυτό θέλησα να αναφερθώ σε αυτό για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μεταρρυθμιστεί η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, διότι είναι δύσκολο ε, να αναγνωρίσει κανείς και να παραδεχθεί ότι ολιγόρησε ότι ήταν αναποτελεσματική η δράση απέναντι στη γρήπη ή τα έναν ή ένα. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μία τετραετία. Το χειμώνα 2009-2010. Ε, νομίζω ότι είναι αρκετά τα προβλήματα αυτά για ένα παγκόσμιο οργανισμό που θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος και να μας καθοδηγεί στην ε, καταπολέμηση αυτού του ιού. Και πολύ σωστά είπατε ότι δυστυχώς μια καταιγίδα ή ε, ένα τυφώνας ήταν, αλλά δεν ήταν μοναδικός ε, ο έμπολα. Θα ακολουθήσουν και άλλοι. Για να συμπληρώσω τα όσα είπε ο αγαπημένος μου συντονιστής Ματίας Γκρότε, θέλω να πω και εγώ ότι συμφωνώ ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να βοηθήσουμε την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για να καταστεί επιτέλους αποτελεσματική. Και ένα τελευταίο συμπερασματικά. Εσείς στη συνεργασία με την ε, ΠΟΗ ε, προετοιμάζετε, εκπονείτε προτάσεις για να μπορεί η διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίζει τέτοιες κατεπίγουσες καταστάσει και κρούσματα. Ας πούμε, τι γίνεται με την αδειοδότηση νέων φαρμάκων, επιταχύνεται η διαδικασία έγκρισής τους. Υπάρχει κανένα πρωτόκολλο. Έχετε σκεφτεί τέτοια ε, συστήματα για να είναι πιο ενισχυμένη και πιο συντονισμένη η απόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Κάντεμπαχ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση και για τη δυνατότητα συζήτησης. Στην παρουσίασή σας μιλήσατε για το πρόγραμμα του τρέχοντος έτους και είπατε, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, ότι επιγόντως πρέπει να πάρουμε επιγόντως μέτρα για την αντίσταση στα αντιβιωτικά, την πολλαπλή αντίσταση. Και επίσης Έχουμε πολλές περιπτώσεις ε, λοιμόξεων στα νοσοκομεία μας. Ήδη με ένα ψήφισμά μας το 2013 το αναφέραμε αυτό. Υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα ήδη για αυτό, αλλά έχουμε τώρα και έναν άλλον σιωπηλό δολοφόνο στα νοσοκομεία μας, το Clostridium difficile, το οποίο δημιουργεί τεράστιες δυσχέρειες. Και τελευταία διάβασα ότι σε 13 κράτη-μέλη υπάρχουν προγράμματα ε, ανείχνευσης αυτού του μικροβίου. Και έχουν αναφερθεί στοιχεία όπως 27.000 ή και περισσότεροι στην Ευρώπη. Ξέρουμε βέβαια ότι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα αντιβιωτικά, άρα, άρα αυξάνεται το ενδεχόμενο περαιτέρω λοιμόξεων και μολύνσεων. Τι θα κάνει ο οργανισμός σας για να αντιμετωπίσει τις νοσοκομιακές ε, λοιμώξεις. Και ιδιαίτερα τη λοιμώξη με αυτό το Clostridium difficile. Τώρα ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή για την παρουσία του εδώ. Επανέρχομαι στα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν για το θέμα της ε, αντοχής, αντίστασης στα αντιβιωτικά και στα αντιμικροβιακά ε, φάρμακα. Είμαι εισηγητής της έκθεσης πρωτοβουλίας ε, η οποία θα πάρει την τελική της μορφή σύντομα. Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω τις εργασίες της υπηρεσίας αυτής ιδιαίτερα στα πλαίσια της παρακολούθησης των λοιμόξεων σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Θίγουν περίπου το 12% των ασθενών σε νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα μέτρα και οι προτάσεις ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Απαιτείται μια σωστή κατάρτιση των, του νοσηλευτικού προσωπικού και των ιδίων των ασθενών εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Ε, μερικές φορές όμως ε, η πολιτική λειτουργεί αρνητικά με την έννοια ότι σε επίπεδο νοσοκομιακό προωθεί κάποια πρόσωπα και κάνει ορισμένους διορισμούς αντίθετα με την έννοια και το κριτήριο της ουσίας και της ποιότητας. Και αυτό είναι κάτι που συνδέεται με δυσάρεστες ε, ε, καταστάσεις. Όταν ένας ιατρός κάνει ένα λάθος διότι δεν έχει τις αρμοδιότητες που πρέπει και τις γνώσεις και έχει διοριστεί για πολιτικούς λόγους, αυτού, του τύπου οι παρεμβάσεις προφανώς είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τους ασθενείς. Δεν ξέρω αν έχει λάβει υπόψη του ο κύριος ε, Διευθυντής ε, τις επιπτώσεις που έχει το φαινόμενο αυτό στην καταπολέμηση των λοιμόξεων σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ευχαριστώ. Τώρα πριν δώσω το λόγο στον ε, προσκεκλημένο μας για να απαντήσει. Να ρωτήσω αν οι εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, οι καθηγητές Μαλιώρη και Σέρες, θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ. Αρχικά να ευχαριστήσω για την ε, εμπιστοσύνη που μου δείχνετε να είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECDC εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, παρακολουθώ τις εργασίες για 10 συνεχή χρόνια. Ειλικρινές ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη σας. Συμπληρωματικά με όσα ακούστηκαν θα ήθελα μόνο να αναφέρω ότι στους επόμενους μήνες θα λάβετε την εξωτερική αξιολόγηση, τη δεύτερη εξωτερική αξιολόγηση που γίνεται βάση του κανονισμού, του ιδρυτικού κανονισμού του κέντρου και έτσι θα έχετε την ευκαιρία, αν διαθέσετε λίγο χρόνο, να δείτε όλες τις δραστηριότητες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και τις συστάσεις ε, εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή των ε, εκπροσώπων των κρατών μελών, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία μέσα από αυτήν την αποτίμηση και την εξωτερική αξιολόγηση να δείτε το σημαντικό ρόλο που παίζει αυτός ο οργανισμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ε, θα ήθελα ε, να εκφράσω την ε, σύμφωνη γνώμη μου και να δω με τα χαράς ότι σημερινό σημείο στην ατζέντα των εργασιών σας είναι λεπτομερή συζήτηση για την κρίση έμπολα, και πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τα συστήματα υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες, διότι πράγματι οι απειλές στη δημόσια υγεία δεν βλέπουν σύνορα, άρα δεν είναι μόνο πώς προστατεύουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά πώς και εφόσον μπορούμε βέβαια, μπορούμε να καλύψουμε και άλλες χώρες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προστατεύσουν τους πολίτες τους, αλλά δυστυχώς, χωρίς να το θέλουν, ίσως επιμολύνουν και πολίτες άλλων χωρών. Ευχαριστώ και πάλι για την σημερινή ε, συμμετοχή μου. Thank you, Professor Sheres. Thank you, Mr. Chairman. Well, as my colleague Mini Maliori, uh, I've been working. Και εγώ, όπως η κυρία Μαλιόρη, ξεκίνησα και δεν κάναμε, είχαμε πρόβλημα, το έκανα, μου Εργάζομαι εδώ και 10 χρόνια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Διευθυντής για τις δραστηριότητες του κέντρου και την ανταπόκρισή μας στις διάφορες χώρες. Όχι ούτε σε αυτά που είπε η συνάδελφός μου κυρία Μαγιόρη για τον ειδικό μας ρόλο ως εκπρόσωπή σας. Χαίρομαι που μπορούμε να παίξουμε αυτό τον ρόλο και ευχαριστώ και όσους σχολιάζουν την έκθεσή μας. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εκπρόσωπό μας ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο, την κυρία Κονέτσνα, με την οποία έχουμε συζητήσει επιμέρους θέματα, καθώς και την συμβολή της κυρίας Κάντεμπαθ και Σρέα για την αντίσταση στα αντιβιωτικά, είναι πολύ χρήσιμη. Την επόμενη περίοδο θα εστιάσουμε κυρίως στην αποτίμηση, να δούμε πού προσφέρουμε θέμενη αξία και η νέα οδηγία για τα, τους διαμεθοριακούς κινδύνους που θέτει σε νέο πλαίσιο τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, ΠΟΗ, εμείς, Κοινοβούλιο, Κομισιόν. Έχουμε παραδείγματα σωστής λειτουργίας αυτού του συσχετισμού. Το θέμα λοιπόν είναι πώς την επόμενη περίοδο θα αντιμετωπίσουμε τις χρηματοδοτικές ε, τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς. Ο ε, επικεφαλής μας εξήγησε ποια μπορεί να είναι τα προβλήματά μας. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή αμέσως πρέπει να σταματήσει ένα μεγάλο τμήμα του προσωπικού μας άλλες ενασχολήσεις για να αντιμετωπίσει μια κρίση όπως τη έμπολα. Άρα το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα που μας υποβάλλονται με βάση τους περιορισμούς. Αυτό έχει να κάνει και με την προσπάθεια αντιμετώπισης της ε, φυματίωσης, έντερο, ε, η το κλωστρίντιουμ. Κάθε στιγμή εμφανίζονται νέες απειλές που θέλουν άμεση παρέμβαση του οργανισμού μας και τροποποιούν ε, το πρόγραμμα εργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εκτελεστικό διευθυντή, ε, τον κύριο Σπρέγγερ, για να απαντήσει. Πόσο χρόνο έχω, δύο λεπτά. Τι δύο. Ε, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε αρκετό χρόνο. Θα ήθελα όμως να σας υποσχεθώ ότι θα επανέλθω και θα σας απαντήσω και γραπτός σε όλες σας τις ερωτήσεις. Ε, προσπαθώ να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κονέτσνα που είναι ο νέος μας σύνδεσμος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας και με έχει εντυπωσιάσει η δράση της, καθώς επίσης και η δέσμευσή της. Αν θέλει να υποστηρίξει ε, χώρες όπως η Μολδαβία, Ουκρανία, η Γεωργία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει πολιτική δέσμευση, το επόμενο βήμα ποιο είναι. Αν μας ζητήσουν εμάς να διαδραματίσουμε ρόλο, πώς να το πω, αυτό δεν θα γίνει μόνο με προσκλήσεις στις ε, συνεδριάσεις μας. Θα πρέπει ουσιαστική να είναι η υποστήριξή μας και αυτό κοστίζει και χρήματα και ανθρωπίνους πόρους, αλλά πραγματικά αυτό χρειάζεται. Πάρα πολύ σημαντικό. Uh, Για τον προϋπολογισμό και τα θέματα των ε, ισοτιμιών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, έχετε δίκιο. Η αγοραστική δύναμη του προϋπολογισμού που παίρνουμε από την Ευρώπη έχει μειωθεί, ενώ αυξάνονται οι ανάγκες και ε, η ζήτηση. Είδαμε τι, γίνεται, τι έγινε με τον έμπολο και δεν είχαμε επιπλέον χρηματοδότηση και είναι καλό να το παρακολουθείτε αυτό. Κύριε Γκρότε, έχετε δίκιο. Έχουμε οδικό χάρτη που ονομάζεται Πολιετές Πρόγραμμα Εργασίες. Έχει ήδη ξεκινήσει για την περίοδο αυτή το 2014. Είναι επταετής η περίοδος και κάθε χρόνο ε, Συμβουλευόμαστε όλα τα κράτη-μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για του συνδέσμου μας και ε, ζητούμε τις προτάσεις σας για το ετήσιο κάθε φορά πρόγραμμα. Και θέλω να σας ε, ευχαριστήσω για τις προτάσεις για το 2016. Περιμένουμε να μας καταθέσετε τις προτάσεις σας. Υπάρχει ακόμα χρόνος συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, διότι είναι πάρα πολλά τα θέματα ε, που μας απασχολούν και τους δύο. Ε, ε, ο όλος τομέας των εμβολίων είναι φυσικά κάτι που αφορά πρώτα τον οργανισμό φαρμάκων από πλευράς φαρμακολογικής και φαρμακευτικής. Από την άλλη όμως υπάρχουν και πολλά θέματα δημόσιας υγείας. Είναι λοιπόν στενή η συνεργασία μας και επίσης ό,τι αφορά το εμβόλιο του έμπολα και έχουμε και κοινά προγράμματα και έργα όπως το IMI ε, και είναι και σε προχωρημένο στάδιο. Είναι πολύ καλή η συνεργασία μας και στενή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία ε, Πύρικ. Βεβαίως ε, ε, ασχολούμαστε και πολύ με τη φυματίωση σε δύο στάδια. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος επιπολασμός φυματίωσης σε κάποιες χώρες. Δεν είναι μεγάλο μυστικό αυτό. Ρουμανία, Βουλγαρία και χώρες Βαλτικής έχουν ιδιαίτερη εμφάνιση φυματίωσης. Αλλά είναι και πολύ ενεργή σε μεγάλες πόλεις. Ο επιπολασμός στο Λονδίνο, στη Ρώμη, στο Ρότερνταμ κτλ. είναι πολύ έντονος. Γι' αυτό Έχουμε μια διτή ε, προσέγγιση απέναντι στη φυματίωση. Ανέφερα και τη Λετωνία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Λετωνία θα διοργανώσει μια συνεδρίαση υψηλού επίπεδου, αν ενθυμούμε καλώ, στις 30 Μαρτίου. Θα συμμετάσχει εκεί και ο οργανισμός μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξ όσων γνωρίζω και ίδιος ο Επίτροπος. Και θα υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στον προγραμματισμό. Να είστε βέβαιοι ότι βεβαίως και μας απασχολεί πολύ η φυματίωση και την παρακολουθούμε. Αναφερθήκατε στις Ηνωμένε Πολιτείε ως προς την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Έχουμε μία κοινή προσέγγιση ε, και προχωρούμε σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης και βεβαίως ε, έχει σημαντικό ρόλο εδώ και η υγεία των ζώων. Γιατί αν υπάρχει μεγάλη χρήση αντιβιωτικών ε, στην κτηνιατρική, αυτό σημαίνει ότι θα αναπτυχθεί πολύ μεγάλη αντίσταση στα αντιβιωτικά στους ανθρώπους. Ε, υπάρχει το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προσέγγιση για την ενιαία υγεία. Συνεργαζόμαστε στενά και με την ΕΦΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ε, σε ό,τι αφορά τις κτηνιατρικές στοιχές και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και για αυτό το θέμα. Θα εκδώσουμε μάλιστα κοινή έκθεση για την αντίσταση ε, στα ε, ε, αντιβιωτικά στα τρόφιμα. Έχετε δίκιο, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στο συντονισμό, στην απόκριση των έμπολα. Έχουμε καλές επαφές με το ΕΚΧΟ, αλλά ίσως στο μέλλον χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε. Κύριε Παρνιό, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικό στο να προβαίνουμε στις συστάσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω καθημερινές επαφές με τους ε, ανθρώπους μας εκεί, επί τόπου. Αν υπάρχει ένα εργαστήριο, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, μπορείς να πας σε μία μέρα ή να είσαι σε μία μέρα απόσταση, ε, ε, καλός, αλλά έχεις αυτοκίνητο. Αν δεν έχεις καύσιμα, τι κάνεις. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που δεν μπορούμε να μπούμε εμεί καν, ε, λόγω ταραχών που επικρατούν εκεί και έτσι έχει πραγματικότητα. Και αυτό δεν μπορεί να λυθεί ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γι' αυτό καλό είναι που υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη, η UNMIR, η ε, πρωτοβουλία εκεί και είναι καλό να υπάρχει μια συνολική αποτίμηση και εκτίμηση του τι πρέπει να βελτιωθεί για να μην ξεσπάσουν και άλλα κρούσματα. Για τον έμπολα είναι θετικά τα νέα, αλλά δεν έχουμε ακόμα πετύχει, κερδίσει τη μάχη. Γνωρίζουμε ότι παραμένει σε απομακρυσμένες περιφέρειες και πώς να το πω. Ε, ε, με την, ναι, με την ε, πρέπει να κατα... με την ευλογιά, συγγνώμη. η ευλογιά έχει εκκριζωθεί, αλλά πρέπει να εκκριζώσεις και το τελευταίο κρούσμα για να είσαι βέβαιος. στον έμπολα ισχύει το ίδιο. Γι' αυτό στη Γουινέα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για την κυρία Κάντενμπαχ. Βεβαίως οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και συμφωνώ. Ιδιαίτερα το Clostridium difficile, το κλωστρίδιο είναι πάρα πολύ ε, δύσκολη περίπτωση και σημαντική. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε, ε, να προωθούμε πρωτόκολλα έτσι ώστε να ανοιχνεύουμε αυτά τα κρούσματα όταν ξεσπούν. Έχω λάβει και μια πρωτοβουλία προσωπικά να δούμε αν μπορούμε να αρχίσουμε μια κατάρτιση για ε, τις ενδονοσοκομιακές ε, λοιμώξεις σε επίπεδο νοσηλευτών. Αλλά γνωρίζετε ότι όταν υπάρχουν τέτοιες λοιμώξεις και, και το, το εντοπίζουν, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης. Σε κάποια νοσοκομεία δεν έχουν ανοιχνευτεί οι λοιμώξεις, όχι επειδή δεν υπάρχουν, αλλά επειδή δεν το γνωρίζουν. Είναι καλό λοιπόν και σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης και να γίνονται συζητήσεις. Εγώ πάντα είμαι υπέρ της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και των στοιχείων για τις ενδοσοκομιακές λοιμώξεις και να δίνουμε και καθοδήγηση αλλά και ε, τους οικονομικούς πόρους που χρειάζονται για την πρόληψη αυτών των παθήσεων. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κύριου Περετσίνη, Δεν έχω ενημέρωση για τις ειδικέ επιτροπές που αναφέρατε για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Μια φορά το μήνα επισκέπτομαι μια χώρα και προσπαθώ να εστιάσω εκεί, προσπαθώ να επισκέπτομαι νοσοκομεία, να συζητώ με τους προέδρους των εκάστοτε επιτροπών για τις ενδοσοκομιακές λοιμώξεις και πολλές φορές εντυπωσιάζομαι. Δεν ξέρω, ίσως επιλέγουν τι μου δείχνουν, Μπορεί, είναι πιθανό και αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα μεταβώ σε ένα νοσοκομείο και ίσως ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα που θίξατε εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως να λειτουργεί σωστά αυτή η Επιτροπή και να παρακολουθεί και να προσέχει. Αυτά. Ε, σύντομα ως απαντήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλες Παρακαλώ. Uh, Όχι, πρέπει να τελειώσουμε γιατί έχουμε υπερβεί και το χρόνο εργασίας των διερμηνέων και νομίζω ότι οι τελευταίοι μίλησαν μόνο αγγλικά, χωρίς διερμηνείς, νομίζω. Αλλά ε, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε το απόγευμα.